σε πράξεις. Εξάλλου είναι καθήκον μας να συμμετέχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα στις ε, συνεδριάσεις αυτής της Επιτροπής και να ενημερώνουμε τα μέλη της Επιτροπής προφορικά ή με γραπτό τρόπο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να διεκπεραιώνουμε τα καθήκοντά μας όσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Βέβαια οι πόροι είναι περιορισμένοι τόσο όσον αφορά εμάς όσο και το Κοινοβουλίο. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να ε, βελτιώσουμε τις μεθόδους εργασίας που χρησιμοποιούμε. Στη Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντος ε, έχουμε οριζόντια προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε θέματα όπως ε, παράνομες χωματερές, μόλυνση της ατμόσφαιρας και κακή διαχείριση υδάτων. Ε, μάλιστα ε, κυρία Πρόεδρε, ο τρόπος με τον οποίο εσείς ε, αντιμετωπίσατε και συμπεριλάβατε τις ε, αναφορές για την προστασία του περιβάλλοντος στη Βουλγαρία είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο επιθυμούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Γιατί ε, τι κάνατε, συγκεντρώσατε όλες τις αναφορές. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι να έχουμε μια περισσότερο πρακτική και στρατηγική προσέγγιση έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να μεγιστοποιήσουμε ε, τις επιδράσεις των πράξεών μας. Ε, το ίδιο πράξατε και εσείς με το να συγκεντρώσετε ε, τόσες πολλές αναφορές. Θα ήθελα εξάλλου να κάνω άλλες δύο προτάσεις που αφορούν στις ε, διαδικασίες ε, της, ε, και τη συνεργασία της δικής μας Γενικής Διεύθυνσης με τη δική σας την Επιτροπή. Εμείς θα χαιρόμασταν αν υπήρχαν τακτικές άτυπες επαφές ανάμεσα στην Επιτροπή σας και τη δική μας τη Γενική Διεύθυνση. Γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε τη διεκπαιρέωση θεμάτων και να βελτιώσουμε τη συνεργασία. Ένα άλλο θέμα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 Sea και κυρίως σε, σε ορεινές περιοχές, κυρίως όσον αφορά τον ε, τουρισμό και άλλες ε, δραστηριότητες. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη Βουλγαρία, παρεμφερεί σε πιέσεις υπάρχουν και σε άλλα κράτη-μέλη και πολύ συχνά έχουμε συζητήσει σε αυτήν την Επιτροπή που αφορούν σε παρεμφερή θέματα κυρίως στη Μεσόγειο. Όμως στη Βουλγαρία υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν σχέση με ελλείψεις ε, της ε, χωροταξίας και έχουν σχέση με την ε, με τον πολλαπλασιασμό μικρών προγραμμάτων που όμως έχουν σωρευτικές επιδράσεις ε, στην ε, ε, φύση. Μία άλλη δυσκολία που υπάρχει είναι ότι πολλά από αυτά τα προγράμματα εφαρμόζονταν ήδη πριν από την ένταξη της χώρας. Ως εκ τούτου τα προγράμματα αυτά δεν υπάγονται στο περιβαλλοντικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, επιθυμώ να ξεκινήσω με κάποιες θετικές παρατηρήσεις. Η εφαρμογή των δύο οδηγιών μας της Natura για τα πτηνά και για ε, τους ε, οικότοπους η ε, ένταξη αυτών των νομοθετικών διατάξεων στο βουλγαρικό δίκαιο εξετάστηκε από την Κομισιόν και δεν διαπιστώσαμε να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή τους. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ σημαντική βελτίωση όσον αφορά την κατάσταση σε σχέση με το 2007. Και θέλω να σας επισημάνω ότι ορισμένες από τις αναφορές ανάγονται πράγματι στο 2007 εξακολουθούν να υπάρχουν ε, κάποιες ε, διατάξεις που θεωρούμε ότι πράγματι ε, δεν εφαρμόζονται. Εμείς λοιπόν συνεργαζόμαστε με τις αρχές της Βουλγαρίας έτσι ώστε να βρούμε την πρέπουσα λύση. Όσον αφορά τον ορισμό των περιοχών του δικτύου Natura 2000 έχει σημειωθεί κάποια βελτίωση το Δεκέμβριο του 2008 εγκρίθηκε ο κατάλογος που είχε κατατεθεί. Η Βουλγαρία καθόρισε τις ε, περιοχές ε, των άγριων πτηνών ως προστατευόμενες περιοχές. Βέβαια, δεν θέλουμε να πούμε ότι όλα βαίνουν καλώς και όλα είναι τέλεια. Συνολικά, πάνω από το 30% του συνόλου της επικράτειας της Βουλγαρίας, δηλαδή πάνω από το 1 τρίτο της επικράτειας της χώρας, σχεδόν διπλασίασε τον αριθμό των προστατευόμενων φυσικών ε, καταφυγίων. Και αυτό σε σχέση με άλλες ε, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι μια θετική είδηση. Τώρα, η αξιολόγηση των ε, επιπτώσεων του δικτύου Natura 2000, για μας αυτό είναι το πιο δύσκολο πρόβλημα. Και θέλω να σας πω ότι είμαστε σε επαφή τόσο με τις αρχές της Βουλγαρίας όσο και με τις ΜΚΟ της Βουλγαρίας για να εντοπίσουμε κάποιες ελλείψεις στο σύστημα αξιολόγησης. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα που πρέπει να συζητηθούν στη συνάντηση που θα λάβει η χώρα τον Οκτώβρη ε, ή τον Νοέμβρη στη Σόφια. Και θα μπορούσε κατά την άποψή μας και ελπίζουμε να ακολουθήσει και ένα άλλο σεμινάριο στις αρχές του 2010. Η ΜΚΟ λοιπόν θα αξιολογηθούν ε, και στις δύο αυτές περιπτώσεις. Όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση, έχουμε δρομολογήσει καλή και αποτελεσματική συνεργασία με τους συναδέλφους μας από τη Γενική Διεύθυνση της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η συγχρηματοδότηση είναι πάντα ένα θέμα που πρέπει να αξιολογείται από τους αρμόδιους οργανισμούς και από την οδηγία Habitat. Η συγχρηματοδότηση επίσης προβλέπεται για την εφαρμογή μέτρων που έχουν άμεση σχέση με την βελτίωση των προστατευόμενων περιοχών στη Βουλγαρία και για τον ε, ορισμό ε, των ε, χώρων που θα μπορούσαν να οριστούν προστατευόμενα καταφύγια. Κάτι άλλο που ενδιαφέρει είναι οι δυνατότητες εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων στην ίδια τη Βουλγαρία. Βεβαίως εφόσον η εφαρμογή γίνεται σε εθνικό επίπεδο και δεν φτάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κατάσταση είναι πάντα καλύτερη. Ένα σεμινάριο για την προστασία της ε, φύσης, για δικαστές πιο συγκεκριμένα, έλαβε χώρα στη Βουλγαρία στο πλαίσιο της ε, δικής μας ε, της οργάνωσης σεμιναρίων για δικαστές που θα ασχολούνται με το περιβαλλοντικό δίκαιο. Αυτή λοιπόν η πρωτοβουλία βοήθησε τους ε, δικαστές στη Βουλγαρία και επίσης ε, τους βοήθησε και στο να εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία. Εξάλλου θέλω να σας πω ότι εξετάζουμε όλες τις ε, διαμαρτυρίες και τις ε, αιτήσει που έχουν σχέση με την κακή εφαρμογή της, προστασίας, της οδηγίας περί προστασίας του περιβάλλοντος στη Βουλγαρία. Πρέπει να πω ότι αυτό δεν είναι κάτι το εύκολο, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει διάδοση, πολλαπλασιασμός μικρών προγραμμάτων και δυσκολίες να διαπιστώσει κανείς κατά πόσον πράγματι εφαρμόζεται το κοινοτικό και το περιβαλλοντικό δίκαιο. Όμως παρόλα αυτά σημειώνουμε πρόοδο. Τώρα, όσον αφορά τον ε, ορισμό των ε, προστατευόμενων ε, οικοτόπων στην Βουλγαρία εντοπίστηκαν κάποιες ελλείψεις όσον αφορά τον ορισμό αυτών των ειδικών χώρων. Εδώ το θέμα που εξετάζουμε έχει σχέση με τα όρια κάποιων ειδικά προστατευόμενων περιοχών. Στην Καλιάτρα εκεί διαπιστώθηκε ε, μία παραβίαση το 2008. Στην περίπτωση αυτή εξετάζουμε το πώς ακριβώς αξιολογήθηκαν η, αξιολογήθηκε ε, η προστασία του περιβάλλοντος και κατά πόσον ελήφθη υπόψη η προστασία αυτής της περιοχής. Πριν από το καλοκαίρι έλαβε χώρα μια επιτόπια επίσκεψη και προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματά της. Στην Κερίν, στο Ήμινε και στο Σάριβο και εκεί υπάρχουν ε, κάποιες ε, έρευνες, συνεχίζονται συνεχίζεται η μελέτη αυτών των περιπτώσεων και θα πρότεινα να επανέλθουμε στο θέμα αυτό κατά την επόμενη συνάντηση της Επιτροπής μας έτσι ώστε να συνεχίσω να μπορέσω να σε ενημερώσω για θέματα και μέτρα τα οποία μεταξύ θα έχει λάβει η Επιτροπή. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις ανησυχίες που έχουν αναφέρει οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί και οι αναφέροντες και επίσης ε, προτιθέμεθα να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε σε μία από τις επόμενες συναντήσεις σας όταν θα έρθει και πάλι το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα λοιπόν, κλείνοντας, να πω και το εξής. Επιθυμώ να επαναλάβω ότι εμείς, η Επιτροπή, οι συνάδελφοί μου ε, από την Επιτροπή Περιβάλλοντο και άλλοι καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία της φύσης στη Βουλγαρία. Γι' αυτό λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, δεν επιθυμώ οι συνάδελφοι της Επιτροπής να κατηγορούνται για κακοδιαχείριση ή για κακή και ανεπαρκή διεκπαιρέωση των καθηκόντων τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Μποτσέλα για την παρέμβασή σας αυτή. Σας ευχαριστώ ε, και για το επικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί είναι πολύ σημαντικό ε, να υπάρχει αυτή η συνεργασία με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να είναι ε, αποτελεσματική ε, η εργασία μας που έχει να κάνει με την προστασία των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Και μην ξεχνάμε ότι αναφέρθηκε και η πρόθεση, ε, μέσα στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος του 2010, αναφέρθηκε ε, και η πρόθεση για διεξαγωγή σεμιναρίων και ε, εδώ πραγματικά είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή στα σεμινάρια αυτά γιατί τα θέματα τα οποία προτίθεστε να συζητήσετε είναι θέματα τα οποία ήδη εμείς από την πρώτη μας συνεδρίαση αναφέραμε και εξετάσαμε. Είναι πολύ ενδιαφέροντα λοιπόν όλα αυτά Τονίζω ότι ε, εμάς μας ενδιαφέρουν τα θέματα αυτά και υπάρχει αυτή η βούληση για συμμετοχή. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο, υπάρχει κάποιος να που το λόγο. Αν δεν θέλει κανείς το λόγο, τότε νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά και πάμε στην επόμενη. Σύμφωνα με αυτά που είπαμε χτες, να δώσουμε δηλαδή προτεραιότητα στις αναφορές όπου παραβρίσκονται, παραβρίσκονται οι αναφέροντες. Πάμε στην 21. Αναφορά 21 λοιπόν. Αναφορά στην οποία είναι παρόν ο Χωσέ Παύλο. Not this one. Όσον αφορά την 21. Uh, Κοιτάξτε, σε αυτά τα οποία είπε η Επιτροπή να προσθέσω το εξή. Εάν η χώρα αλλάξει τα έργα, Ε, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν θέλω να πω, επειδή τα άλλαξαν, αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται για κοινοτική χρηματοδότηση και πλέον δεν ασχολούμαστε με αυτά. Με εξέπληξε κάπω αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία, ευχαριστούμε. Να πάμε στο 21. Πέτρο Χιμένε. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και επιτρέψτε μου σήμερα να ε, σας μιλήσω για το θέμα αυτό. Θέλω να μεταφέρω μια πλατφόρμα των πολιτών που δημιουργήθηκε το 2002 και που αποτελείται πάνω από 30 οργανώσεις των πολιτών, ενώσεις, ε, και, αλλά και πολυάριθμα άτομα, τα οποία σε προσωπική βάση ανήκουν σε αυτή την πλατφόρμα. Ε, η πλατφόρμα ε, ε, ασχολείται με το Δέλτα του Γουέλβα και στην οποία συμμετέχει και η δική μου η πολιτική ομάδα και 25.000 άτομα από το Μάιο στο Νοέμβριο του 2008 υπέγραψαν την αναφορά που έχετε μπροστά σας σήμερα και που εξετάζεστε. Κύριε Πρόεδρε, στην Ουέλβα στη δεκαετία του 1960 ε, υπήρξε, ε, υπήρξε μια σειρά από βιομηχανικέ εγκαταστάσει που διαβρίθηκαν με την πάροδο του χρόνου μέχρι να φτάσουμε στη σημερινή του μορφή. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε ένα βιομηχανικό πάρκο με ισχυρή συγκέντρωση χημικών εργοστασίων, ε, ε, θερμικών εργοστασίων, διηληστήρια τα οποία βρίσκονται στο στάδιο διεύρυνση αυτή τη στιγμή και μια τρομερή συγκέντρωση αποθεμάτων αερίου που πραγματικά έκαναν την περιοχή αυτή ε, βασική ε, περιοχή αποθέματος αερίου. Λοιπόν, ε, όλα αυτά βρίσκονται φαινός μέσα στην Ουέλβα και, φετε, φετέρου στην ε, Πάλοντε Λαφροντέρα που είναι, που είναι η διπλανή περιοχή. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι από τις βιομηχανίες που βρίσκονται στο βιομηχανικό πάρκο της Ουέλβα μόνο η Φερτιβέρια ΕΣΕΑ αυτή τη στιγμή καλύπτει 1.200 εκτάρια δημόσιας γης. Ε, στην, σε, μια σε μια περιοχή ε, κοντά στο, ποτάμι, στο ποταμό Τίντο. όσον αφορά την περιοχή αυτή πρέπει να πούμε ότι σήμερα υπάρχουν πάνω από 120 ε, εκατομμύρια τόνοι φωσφογύψου. Μιλάμε λοιπόν ε, για ε, βιομηχανικά απόβλητα τα οποία βρίσκονται σε 500 μέτρα από την αστική περιοχή. Όσον αφορά το φωσφογύψο, ε, εκτός από αυτό υπάρχουν και 7.000 ε, τόνοι ε, ραδιοενεργούς στάχτης λόγω ενός ατυχήματος που έγινε στο Κάντις. Λοιπόν, απέναντι σε ολόκληρη αυτή την κατάσταση είναι ουσιαστική σημασίας η Επιτροπή Έρευνας ε, που ενεκρίθη τότε από την Επιτροπή Αναφορών και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για το σκοπό αυτό. Πρέπει λοιπόν η διερευνητική αυτή Επιτροπή να πάει στον δόν πιο σύντομα ε, στην Ουέλβα για να δει επιτόπου την κατάσταση περιβαλλοντικής επιδείνωσης και ε, ε, τις επιπτώσεις που έχει όλη αυτή η βιομηχανική δραστηριότητα στην πόλη Βέλβα. Ταυτόχρονα ε, είναι απαραίτητο να, σταματήσει, να σταματήσουν αυτά τα απόβλητα φωσφογύψου άμεσα. Γιατί μετά από τόσο χρόνο που πέρασε, από τότε δηλαδή που η Γενική Διεύθυνση Ακτών που εξαρτάται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος είχε αποφασίσει να σταματήσει αυτή η κατάσταση, ταυτόχρονα αυτή η συγκεκριμένη επιχείρηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου 2012 επιτρέπεται να ρίχνει τα απόβλητα αυτά. Και μάλιστα χτες ε, που ήταν η μέρα συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών ε, πρέπει να πω ότι δημοσιεύθηκε στην Ισπανία το γεγονός ότι Ακριβώ πρέπει είχε πάρει αυτή την παράταση μέχρι την 21η Δεκεμβρίου του 2012 όπου θα εξακολουθεί ε, να ρίχνει τα αποθέματα φωσφογύψου ή ε, ε, το εργοστάσιο αυτό. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η δραστηριότητα και να καθαρίσει η περιοχή μετά από αυτή τη δραστηριότητα των 40 ετών ενώ θα πρέπει ταυτόχρονα αφού θα πάψει αυτή η βιομηχανική δραστηριότητα που δεν πρέπει να συνεχίσει να δοθούν εναλλακτικέ λύσει στους εργαζόμενου. Επίση, όσον αφορά αυτέ τι 7.000 ε, τόνου ε, ε, ραδιενεργού στάχτη, πρέπει να μεταφερθεί σε ένα ασφαλή τόπο, ο οποίο να είναι προορισμένο για αυτά τα συγκεκριμένα επικίνδυνα απόβλητα. Πρέπει να σα πω, κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, ότι οι πολίτε έχουν μεγάλε προσδοκίε και περιμένουν πολλά από την απόφαση τη Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφορών, διότι στο τέλο προηγούμενη θητεία ενεκρίθη η δημιουργία αυτή τη Διερευνητική Επιτροπή που θα μεταφερθεί μεταβεί στην Ουέλβα και αυτό το οποίο επιθυμώ είναι η επίσκεψη αυτή να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ γιατί ε, συγκεκριμενοποιήθηκε στην συνεδρία των συντονιστών η επίσκεψη αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. David Hammerstein. Καλημέρα σας σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την Πρόεδρο ε, της Επιτροπής. Αυτή τη στιγμή ε, βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας δύο αναφέροντες, τον εκπρόσωπο της Greenpeace Ισπανίας και την οργάνωση μέσα δελαδρία de Huelva ε, της οργάνωσης που είναι μια που, που, δημιουργήθηκε νόμιμα ακριβώς για το σκοπό αυτό για, την, για τον καθαρισμό της περιοχής ε, κοιτάξτε, μιλάμε για το πιο, ίσως για το πιο ε, σημαντικό ε, χώρο, ρηπογόνο χώρο της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κατάφορη παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Η Ισπανική κυβέρνηση όμως είπε τώρα θα δώσει άλλα 3,5 χρόνια ε, περιθώριο στην βιομηχανία αυτή. Μάλιστα. Από τη μια μπορεί να πει κανεί ότι είναι μια πρόοδος. Από την άλλη όμως μιλάμε για κατάφορη γελιοποίηση του ευρωπαϊκού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα ε, κράτησε ιδιαίτερα παθητική και αργή δράση. Έστειλε επιστολή προειδοποιητική, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που αποτελεί ε, κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και παραβιάζει την οδηγία για τα τοξικά απόβλητα, ε, την οδηγία για τι χωματερέ και εδώ μιλάμε και για μια ζώνη του Natura 2000. Ε, ε, που είναι ακριβώ γιατί και εκεί ε, μιλάμε για τον ποταμό αυτό όπου έχουμε βαρέα μέταλλα και ραδιενεργείς ουσίες. Κοιτάξτε, πρέπει να σα πω ότι ε, με την προεδρική Επιτροπή δεν λύνεται τίποτα. Ε, επιστολή δεν, δεν έγινε τίποτα. Με τι προειδοποίησει τίποτα δεν γίνεται. Τώρα πρέπει να έχουμε ε, συγκεκριμένη αποκατάσταση τη περιοχή. Μιλούμε για, μια ε, για, για ένα σκάνδαλο. Ε, απάτη, ψεύδι, για μια παράνομη δραστηριότητα που γίνεται εδώ και δεκαετίε. Η άδεια αφορά τρία μέτρα αποβλήτων. Αλλά σήμερα έχουμε 30 μέτρα. εάν, κοιτάξτε, Μελετάται μελετάτε η περίπτωση αυτή ε, από όλου ε, όλους όσους ασχολούνται με τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο. Από το Πανεπιστήμιο Πομπέους Φαύρα, από το Πανεπιστήμιο Κάρλος Τερθέρο της Ισπανίας υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες για τις σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία η Ουέλβα ε, έχει τα υψηλότερα ε, κρούσματα, ε, από τα υψηλότερα κρούσματα ασθματικών. Στην πέμπτη, στην έκτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Καρκίνος του πάνω από 15% από την υπόλοιπη Ισπανία. Μιλάμε για ένα σοβαρότατο πρόβλημα το οποίο απαιτεί άμεση απάντηση. Απευθύνω έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στείλτε αιτιολογημένη γνώμη φέρτε την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί πραγματικά δεν πρέπει να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Τι, τι πρέπει να γίνει. Δημιουργήθηκε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων στην Ουέλβα και ε, πραγματικά ε, η, η, επιτροπή αυτή στερείται αξιοπρεπίας. Γιατί, γιατί οι επικεφαλείς είναι αυτοί που υποστήριζαν ε, τη βιομηχανία. Ε, υπάρχουν επιστήμονε εκεί που λένε ότι δεν υπάρχει ε, κανένα κίνδυνο στη δημόσια υγεία. Ο κύριο Ολίβα, για παράδειγμα. Και ε, αποκλείστηκε οποιοδήποτε επιστήμονας, οποιοδήποτε άνθρωπος ε, που γνωρίζει τι έγινε, αποκλείστηκαν οι αγωνιστές αυτοί που προσπάθησαν να καθαρίσουν την περιοχή. Η Greenpeace ζήτησε να αποστείλει σε αυτή την Επιτροπή τεχνικούς εμπειρογνώμονε. και ε, η τοπική κυβέρνηση Ανδαλουσίας απέκλεισε αυτή την περίπτωση. Κανείς εκπρόσωπος των πολιτών, κανείς επιστήμονας που έχει αντίθετη άποψη δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή την Επιτροπή. Μιλάμε λοιπόν για αναξιόπιστες προσπάθειες. Ε, μιλούν ε, για φύτευση δέντρων, μιλούν ε, για αποξήρανση περιοχής, μα δεν μιλούν για αφαίρεση των βαρέων μετάλλων, ε, των ραδιενεργών στοιχείων. Φοβάμαι λοιπόν ότι εδώ πρόκειται για ένα τρομερό κενό. Δεν, δεν, δεν πρέπει να σταματήσουν μόνο οι απορρίψεις, αλλά πρέπει να γίνει και η επεξεργασία των αποβλήτων. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν, να υπάρξει απόλυτη συμμόρφωση, πλήρη συμμόρφωση με την νομοθεσία από την επιχείρηση αυτή. Γιατί η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι ε, ε, εφαρμόζεται η αρχή ο πληρώνει. Αυτό που μας απασχολεί σε σχέση με την κυβέρνηση Ανταλουσίας αυτή τη στιγμή είναι ότι από ό,τι φαίνεται, αυτά θα τα πληρώσουν οι Ισπανοί φορολογούμενοι και ενδεχομένω και οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι και όχι αυτοί που προκάλεσαν τη ρήπανση αυτή. Και κάτι άλλο. Όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, θα πρέπει να γίνει, η επεξεργασία των αποβλήτων θα πρέπει να γίνει με όλε τι περιβαλλοντικέ εγγύησει. Ζητώ από την Επιτροπή να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μα. Όχι μόνο επίσκεψη πολιτική φύσεω, αλλά ε, ε, να υπάρξει αμερόληπτη επιστημονική ε, μελέτη ε, γιατί αυτό δεν το επέτρεψε ε, η, τοπική κυβέρνηση Ταλουσίας η οποία προσπάθησε να κουκουλώσει το ζήτημα. Έφτιαξε την επιτροπή σα είπα που υπάρχουν επιστήμονε που μιλούν για έλλειψη κινδύνου. Εδώ μιλάμε όμως για απόβλητα ε, και ε, για κατάλοιπα. Δεν μιλάμε για υποπροϊόντα. Μιλάμε για κατάλοιπα, για απόβλητα επικίνδυνα και έχουμε παραβίαση συγκεκριμένη νομοθεσία. Ζητάμε τη ε, συμμετοχή περιβαλλοντικών οργανώσεων όπως Μέσα Δελαρία, ε, Greenpeace ε, στην Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα ε, αποφασίσει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Απαιτούμε επιστημονική αξιολόγηση για όλη τη ζώνη, συμπεριλαμβάνοντας και τον ποταμό. Η, ζώνη βρίσκεται στη, στο Natura 2000, στο δίκτυο Natura 2000 και μιλάμε για βαρέα μέταλλα, για ραδιενεργείς ουσίες. με δύο λόγια ζητάμε άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Να σας πω και εγώ κάτι. Η συνεδρίαση των συντονιστών ε, μόλις συμφώνησε ότι θα γίνει επίσκεψη στην ΟΕΛΒΑ. Η Γιολάντα Βιλάρη, εκπρόσωπος Κομισιόν, θα μιλήσει τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ που μα ε, καλέσατε να τοποθετηθούμε εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμμετάσχουμε στη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ του αναφέροντε και του εκπροσώπου των αναφερόντων για αυτή την παρουσίαση του θέματο. Πράγματι, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ε, το γνωρίζει η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι συνηθισμένο το θέμα αυτό, ε, με την έννοια ότι εξετάζεται αρκετέ φορέ στην Επιτροπή Αναφορών. Και θα ήθελα να πω ότι εμεί παρακολουθούμε με επίγνωση του επίγοντος χαρακτήρα το ζήτημα. Έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα ότι εδώ πρόκειται για ένα πρόβλημα περιβαλλοντικής φύσεως το οποίο πρέπει να εξεταστεί με τη δέουσα προσοχή και να δούμε τη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο. Το μόνο που θέλω να πω ε, είναι να μιλήσω για το περιβαλλοντολογικό δίκαιο και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στο συναδελφό μου, ε, τον κύριο ε, Μάσιμο Αρίμπα, εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, ε, για να ενημερώσει τους αναφέροντες για την ε, πιθανή παραβίαση της οδηγίας 96-26 ευρωτών που αναφέρεται στις πιθανές επιπτώσεις των εργαζομένων ε, στους εργαζόμενους και στους ε, πολίτες από αυτές τις ραδιενεργικέ ουσίες. Θέμα στο οποίο αναφέρθηκαν και διάφοροι αναφέροντες. Δηλαδή στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία πρόκειται για μία βιομηχανική δραστηριότητα που συνεπάγεται την αναπόθεση φωσφογύψου και βεβαίως όλα αυτά είναι ραδιενεργά υλικά ε, ταυτόχρονα έχουμε ε, και την, ε, αυτές τις στάχτες που περιέχουν διάφορες ρενεργικές ουσίες και κυρίως κέσιο 137. Θα ήθελα λοιπόν να ε, ενημερωθείτε για, τα τελευταία στοιχεία. Όσον αφορά λοιπόν την παραβίαση του περιβαλλοντολογικού δικαίου ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, έχει γίνει ενημέρωση τακτά χρονικά διαστήματα ε, για το τι έχει γίνει στο ζήτημα αυτό. Νομίζω η τελευταία παρέμβαση επιτροπής ήταν τον Απρίλιο αυτού του έτους ε, και στο μεταξύ Α, να σας περιγράψω, να σας μιλήσω για τα βασικά χρονικά σημεία, για τα βασικά ορόσημα και να σας πω τι έχει γίνει. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ε, προσφυγής κατά των δύο αυτών ε, εργοστασίων που βρίσκονται στο βιομηχανικό πάρκο ε, της Ουέλβα ενημερώθηκε για το ότι ρίχνουν τα ε, λεγόμενα απόβλητα φωσφογύψου που προέρχονται από τη βιομηχανική ε, διαδικασία παρασκευή λιπασμάτων σε συγκεκριμένη περιοχή. Πρέπει να πούμε και αυτό εξ αρχή, ευθύ εξ αρχή, ότι η, αυτή η δραστηριότητα όπως, όπως είπε και ο αναφέρον, δεν, δεν είναι κάτι που ξεκίνησε πρόσφατα. Πρέπει λοιπόν να θυμίσουμε ότι οι δραστηριότητες εναπόθεση του φωσφογύψου άρχισαν ήδη από τη δεκαετία του 60, ε, τη στιγμή που ε, ιδρύθηκε αυτό το βιομηχανικό πάρκο. Και επομένως ε, τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να εξετάσει την νομιμότητα δράσεων που προηγήθηκαν τις ε, θέσεις ε, σε ισχύ του κοινωτικού δικαίου. Μιλάμε λοιπόν για το γεγονός ότι πρέπει τώρα αυτή τη στιγμή ε, να ε, ανακτηθεί μια περιοχή ε, που υπέστη αυτή την αντιμετώπιση εδώ και τόσα χρόνια. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να το καταλάβουμε όλοι ότι εδώ οι συγκεκριμένες δραστηριότητες ξεκίνησαν πριν την θέση σε ισχύ των οδηγιών. Βεβαίως είναι απόλυτα νόμιμο ε, οι πολίτε να ζητούν την ανάκτηση τη περιοχή του, αλλά αυτή τη στιγμή εξετάζουμε την εφαρμογή των υποχρεώσεων του κοινοτικού δικαίου και δεν μπορούμε ε, να ε, αναφερθούμε σε δραστηριότητε που ανέρχονται στη δεκαετία του 60, όπου ούτε καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, βρισκό, δεν η Ισπανία. Και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για εφαρμογή οδηγιών που εφαρμόζονται τώρα. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Και βεβαίω με την επιφύλαξη όλων αυτών θα ήθελα να προχωρήσω στην ανάλυση της υπόθεσης. Πιστεύουμε ότι οι δραστηριότητες αυτών των δύο καταστάσεων πρέπει ε, να, ε, να συμφωνούν με την οδηγία η οποία αναφέρεται στον έλεγχο των εκπομπών ε, IPPC και να δούμε τι γίνεται με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι όταν ήρθαμε σε επαφή με τις αρχές ε, για να δούμε ε, κατά πόσον έχουν δοθεί συγκεκριμένε άδειε ε, που να προβλέπουν, που να προβλέπουν τις ορισμένες δικλείδες ασφαλείας. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν οι άδειε αυτές. Στείλαμε λοιπόν επιστολή και στη συνέχεια, το 2008, στη συνέχεια οι αρμόδιες αρχές προέβησαν σε εγκρίσεις IPPC τον Απρίλιο του 2008 ε, μετά από τη δική μας την προειδοποιητική επιστολή και τότε εμείς αρχίσαμε να εξετάζουμε τις προϋποθέσεις ε, που λαμβάνονται για τις ε, ρήψεις φωσφογύψου για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και για αυτό το λόγο πραγματοποίησαμε επίσκεψη επιτόπου ε, που είναι κάτι το οποίο γίνεται εξαιρετικά, σε εξαιρετικέ περιπτώσει. Και γι' αυτό θα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι πήραμε πολύ σοβαρά την υπόθεση αυτή και θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητο να δούμε επί τόπου τι ακριβώ γίνεται ε, και πώ έχουν τα πράγματα όσον αφορά ε, αυτά τα απόβλητα και αυτά όλα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη ε, κατά την αξιολόγηση ε, της ε, κατάστασης. Ε, γι' αυτό ε, ήσαμε επιτόπου με τις αρχές αυτές για να δούμε τι γίνεται ε, και να μην ε, στηριζόμαστε σε κάποια απλά έγγραφα τα οποία μπορεί να μην δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει να σας πούμε ότι μετά από την επίσκεψη αυτή τον Νοέμβριο 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε τις, ε, ε, τι, ε, τι γίνεται και στείλαμε εξυπηρετική επιστολή για να ξεκινήσουμε εκ νέου τη διαδικασία, ζητώντα από τι αρχές να εφαρμόσουν, ε, να, να συμμορφωθούν με τι υποχρεώσει ε, που απορρέουν από την οδηγία. Προς την κατεύθυνση αυτή λοιπόν, και όπως ακριβώς αναφέρθηκε από τον κύριο Χάμερστριτ, να, να, να επιβεβαιώσω και εγώ ότι η Επιτροπή θεώρησε ότι ο φωσφογύψος Ε, μπορεί να είναι και υποπροϊόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ε, απόβλητο, δεν είναι κατάλοιπο. Ε, θεωρείται και ως κατάλοιπο, άρα λοιπόν πρέπει να θεωρήσουμε ότι στις πιζώνες αυτές γίνονται απορρίψεις αποβλήτων. Με την έννοια αυτή, η οδηγία IPPC μαζί με την συγκεκριμένη οδηγία που αφορά τις απορρίψεις είναι οι οδηγίες που θα πρέπει να εφαρμοστούν και που θα πρέπει να πληρούν οι αρμόδιες αρχές. Αυτά τα νομικά ζητήματα λοιπόν, τα νομικά επιχειρήματα αναφέρθηκαν στις Ισπανικές Αρχές και όπως σας είπα προσπαθήσαμε να δούμε πώς ακριβώς εφαρμόζονται συγκεκριμένε οδηγίες ε, στην περίπτωση αυτή ένα απόρριψη του φωσφογύψου και αυτή τη στιγμή εξελογούμε την απάντηση της, ε, των Ισπανικών Αρχών που εδώ το 2009. Όπως τόνισαν, ε, όπως τόνισε και ο Χάμερ Σμιθ, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο ε, ε, ζήτημα, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το τεχνικό πρόβλημα. Δεν είναι θέμα κατά πόσον πρόκειται για απόβλητα ή όχι. Εμεί είπαμε ότι πρόκειται για απόβλητα, αλλά το θέμα είναι να δούμε κατά πόσον ε, εφαρμόζουν σωστά την οδηγία για τα απόβλητα και την οδηγία IPPC και να δούμε ε, κατά πόσον ε, οι συγκεκριμένες, ε, η συγκεκριμένη απόρριψη αποβλήτων δημιουργεί προβλήματα στην υγεία. Εξετάζουμε λοιπόν λεπτομερώς και εμπεριστατωμένα όλες αυτές τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες τεχνικού χαρακτήρα. Αλλά αυτή τη στιγμή ακόμα δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Όπω είπα, είναι πολύ μπλοκό το ζήτημα και ακριβώ γι' αυτό δεν έχει ληφθεί απόφαση από τι διαδικασίε. Πάντω, θα ήθελα να επαναλάβω τη δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσουμε την, ε, ε, την εμπεριστατωμένη μελέτη ε, όλων των στοιχείων ε, που θα πρέπει να πληρούνται για την απόρριψη φωσφογύψου ε, τονίζουμε ότι πρόκειται για 1.200 τόνου φωσφογύψου. Θα ήταν δεν θα ήταν δυνατόν να μεταφερθούν σε άλλη περιοχή. Απλά και μόνο πρέπει να δούμε κατά πόσον εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις ε, στα, στις υφιστάμενες που χρησιμοποιούνται ως περιοχές ε, απόρριψης αποπλήτων. Σχετικά σύντομα ελπίζουμε να έχουμε καταλήξει σε μία απόφαση και αυτό που θέλουμε είναι να εξασφαλίσουμε την συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο όσο δυνατόν πιο γρήγορα και όσο το δυνατόν ε, πιο ε, θετικά και υπέρ των πολιτών. Να δώσω το λόγο στον συνάδελφο της ε, Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για τα θέματα που αφορούν στη ραδιενέργεια και στα απόβλητα σε αυτήν την αναφορά. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να σας πω ότι την κύρια ευθύνη για τον έλεγχο των επιπέδων ραδιενέργειας ε, που ε, προκύπτουν από τέτοιου είδους αναπόθεση αποβλήτων, η κύρια ευθύνη βρίσκεται στα χέρια των εθνικών αρχών. Η Κομισιόν αυτό που κάνει είναι να ελέγχει τις ε, εγκαταστάσεις ε, ελέγχου ραδιενέργειας και κατά πόσον οι μετατροπές που είναι απαραίτητες εφαρμόζονται σωστά από τις εθνικές αρχές. Πέρα από αυτό που ανέφερε η Κομισιόν κατά τη τελευταία μας συνάντηση τον Απρίλιο όταν συζητήθηκε αυτή η αναφορά, λάβαμε και μία σειρά αναφορών από διάφορες αρχές στην Ισπανία και επίσης και από τους ε, ίδιους τους ε, αναφέροντες. Πιο συγκεκριμένα λάβαμε μία ε, αναφορά από την Conseil National και από, την, από το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων μία έκθεση επίσης από ΜΚΟ και όλες αυτές οι εκθέσεις αναλύθηκαν από, τους, από τα στελέχη της Κομισιόν. Τώρα, όσον αφορά την ε, έκκληση των, ε, την ραδιενεργη συγκεντρωση συγκέντρωση CS137 η έκθεση αναφέρει ότι πράγματι ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια που προβλέπονται στην Οδηγία 96-29 σχετικά με ε, την ακτινοβολία από Εκεί υπάρχουν διαφορετικά όρια έκθεσης και εδώ μοιάζει να υπάρχει κάποια αντίφαση. Με πάση περιπτώσει, η Κομισιόν γνωρίζεται πολύ καλά πόσο περίπλοκο είναι το θέμα. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να ε, έχουμε μια αποστολή επιτόπου που θα κάνει τον έλεγχο μια αποστολή της Ευρατόμ και η οποία θα ελέγξει ότι οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν το μηχανισμό ελέγχου που χρησιμοποιείται από τις ισπανικές αρχές ε, πράγματι λειτουργεί σωστά. Αυτή λοιπόν η αποστολή θα λάβει χώρα το φθινόπωρο αυτού του έτους και εγώ θα σας ε, αναφέρω, θα επανέλθω στην Επιτροπή και θα σας ενημερώσω μετά από το πέρας αυτής της ε, αποστολής. Ευχαριστώ. Θέλει κανένα να, πάρει, να παρέμβει παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους αναφέροντες, ιδιαίτερα ε, τον εκπρόσωπο της πλατφόρμας, γιατί έχει ε, φέρνει μαζί του 25.000 υπογραφέ των πολιτών ε, της Γουέλβα που εξέφρασαν την ανησυχία τους, Συνοδεύοντα την αναφορά αυτή. Κοιτάξτε, το θέμα αυτό το συζητήσαμε σε βάθος την προηγούμενη θητεία. Θυμάμαι ε, την παρουσία δύο αναφερόντων από την Greenpeace και τον κύριο Βασίλια και πρέπει να σας πω ότι η συζήτηση έγινε σε βάθος και καταλήξαμε με την συμφωνία μας, ε, τη συμφωνία όλων μας, να στείλουμε αποστολή. Ε, αναβλήθηκε η επίσκεψη αυτή λόγω των ε, ευρωπαϊκών εκλογών και συμφωνήθηκε μετά τις εκλογές να στείλουμε αυτή την διερευνητική επιτροπή ε, στην ΟΕΡΒΑ. Χαίρομαι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που όπως ακούσαμε από την εκπρόσωπό της ε, δεν είναι ε, κάτι το οποίο συνηθίζεται. Χαίρομαι γιατί αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάει στην Ουέλβα. όπως και οι πρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας που κατέληξαν στη συμφωνία να επισκεφθούν την ΟΕΛΒΑ, γιατί είναι κρίσιμη σημασία στο θέμα αυτό. Έχει να κάνει με ε, ραδιενέργεια ε, και, με, και χαίρομαι γιατί σήμερα το πρωί ε, στη συνεδρία των συντονιστών ομόφωνα αποφασίστηκε να ε, συγκεκριμενοποιήσουμε την απόφαση της Επιτροπής Αναφορών και να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας. Να πάμε στην Ουέλβα, να έρθουμε σε επαφή με τις αρχές, η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας θα κάνει το ίδιο. Λοιπόν, και εμείς πρέπει να δράσουμε σύντομα. Έτσι ώστε πράγματι, όπως ε, είπε και πολύ σωστά χτες ο σύντροφος Μαρτίνες, όταν μιλούσαμε για τη Σεβίλη, ναι, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει υλικό ε, υπάρχει ε, ε, λόγος να παρέμβει η Επιτροπή και να πάει στην Σεβίλη, όχι έχοντας αποφασίσει εκ των προτέρων θα κάνουμε και προδικάζοντας τα πράγματα, να έρθουμε σε επαφή με όλες τις πλευρές. Γιατί νομίζω ότι οι αρχές της Ανταλουσίας είναι προς το συμφέρον τους να ξεκαθαρίσουν το εξής. Τι θα γίνει πρώτα απ' όλα με αυτούς 125.000 τόνους φωσογύψου που καλύπτουν επιφάνεια, ε, ίδια με την επιφάνεια τη ε, πρωτεύουσα Χουέλβα. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε το ερώτημα στην επιστημονική κοινότητα. Τι θα γίνει με αυτού του τόνου. Και δεύτερον, όσον αφορά το επίπεδο ραδιενέργεια. Να σα πω το εξή. Εγώ πήγα με έναν πυρογνώμονα σε θέματα ραδιενέργεια. Πήγα, πήγα, εκεί. Με έναν πυρογνώμονα που είχε μετρητή Γκάγκερ. Που όπω ξέρετε, ο μετρητή Γκάγκερ μετρά την ακτινοβολία. Εγώ πήγα φορώντα ειδική στολή. Ε, όπω καταλαβαίνετε, και εγώ διάλεξα προσωπικά τρεις διαφορετικές ε, περιοχές από την ε, υγειονομική ταφή του φωσφογύψου. Με εκεκριμένο μετρητή Γκάιγκερ μέτρησε ο εμπειρογνώμονας ε, πάνω από 400 φορές, περισσότερο από το όριο που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν κυρία Πρόεδρε ότι βρισκόμαστε απέναντι σε μια κατάσταση που δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει κανείς για δημαγωγικούς σκοπούς. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Νομίζω λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί, να μην ε, κινδυνολογήσουμε άσκοπα και δημιουργήσουμε πανικό, αλλά όπως κάναμε ήδη, να δώσουμε συγκεκριμένη ημερομηνία επίσκεψη και να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και να υποβάλει έκθεση η διευρυντική Επιτροπή στην Ολομέλεια τη Επιτροπής μας. Στη συνεδρίαση των ε, συντονιστών είχαμε πει ότι το κάθε μέλος ε, δεν πρέπει να μιλάει, δηλαδή ο κάθε βουλευτής δεν πρέπει να μιλάει πάνω από 2-3 λεφτά το πολύ. Σας παρακαλώ μην με αναγκάζετε να σας διακόπτω, γιατί αλλιώς ε, τι νόημα έχει. Αν εμείς ήδη δεν σεβόμαστε ας πούμε τους, τις δεσμεύσεις μας, δεν θα σεβαστούμε καμία άλλη. Ποια άλλη δέσμευση μπορούμε να σεβαστούμε. Ε, αυτά που παίρνουμε, τι δεσμεύσει που αναλαμβάνουμε για, τους επισκέπτε, για τις επισκέψεις κτλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε δύο-τρία λεπτά να ολοκληρώσουμε τι απόψει μα για το θέμα αυτό. Κοιτάξτε, όσον αφορά το θέμα αυτό, υπάρχουν πολλά στοιχεία που μα βρίσκουν όλου σύμφωνου. Πολύ συνοπτικά το λέω. Πρώτον, ότι έγιναν απορρίψεις ε, που προκάλεσαν σοβαρή ρήπανση και της περιοχής και το, του ποταμού Τίντο. Δεύτερον, ότι οι δημόσιες αρχές ε, εδώ και 20 χρόνια ασκούν πίεση στα δύο αυτά εργοστάσια έτσι ώστε να αλλάξουν το σύστημα απόρριψης που ε, ε, ε ακολουθεί τώρα ένα, ένα κλειστό κύκλωμα υδατός αλλά παρόλα αυτά και παρόλα στις νέες εγκαταστάσεις ε, γιατί κοιτάξτε, υπάρχει και τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου. Ε, δεν μπορεί κανεί. Ε, ε, ε Βέβαια, πρέπει να καταλάβουμε ότι ε, το εργοστάσιο δεν κλείνει μια μέρα στην άλλη. Έτσι. Ε, δόθη λοιπόν προθεσμία μέχρι το 2012. Τώρα, ε, είχε δοθεί η αρχική άδεια μέχρι το 2007. Τώρα, ε, ήδη έχει κλείσει το 50% των εγκαταστάσεων αυτών απόρριψη και μέχρι το 2012 έχει προθεσμία για να τι κλείσει όλε. Από ό,τι έχω καταλάβει, δεν υπήρξε κανένα είδο απειλή στην ανθρώπινη υγεία. Ούτε καν ελάχιστη φύσεω. Ούτε δερματικά προβλήματα, ούτε άσθμα, ε, ούτε καρκίνο. Το Πανεπιστήμιο τη Σεβίλη, τη Μάλαγα, τη ε, ε, της Βουέλβα, το, το Συμβούλιο Πυρηνική Ασφάλεια είπε ότι δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο. Βεβαίω. Εγώ δεν μπορώ να σα το πω ξεκάθαρα, βέβαια. βέβαια. Καταλαβαίνω πολύ καλά και αυτά τα οποία είπε ο κύριο Μπίλι Μάγερ. Να δούμε τι θα κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα τελειώσει τώρα στο φθινόπωρο και στη συνέχεια μπορούμε να έχουμε ε, αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αποστολή έτσι, όχι διερευνητικής φύσεως Ε, η οργάνωση μέσα στα βελαρία και ο κύριος Βίλι Μέγερ θα καταλάβει ότι ταυτόχρονα ε, έχουμε ε, τόσους εργαζόμενους και που έχουν άμεση εργασία και έμεση. και εδώ μιλάμε για την Ούχετε και την Κομισιόν Εσομπρέρα στα δύο μεγάλα συνδικάτα, τα οποία διαφωνούν με το κλείσιμο των εργοστασίων. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Πάντω, εγώ να σα πω, εγώ προσωπικά, αλλά και το κόμμα μου και οι, οι, οι δημόσιε αρχέ πιστεύουν πρέπει να κλείσουν τα δύο αυτά εργοστάσια. Τέλο. Πιστεύω, προτείνω, αλλά βεβαίω εσεί αποφασίζετε. Πιστεύω ότι η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών πρέπει να πάει αφού ε, γίνουν γνωστές οι μελέτες βρατόμ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τουργκάης. Ε, Ευχαριστώ. Εδώ μιλάμε... Εδώ μιλούσαμε για, το ποια, για ποια επιτροπή μιλάμε, την Επιτροπή τη δική μα ή την, επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε, χθες ε, όσον αφορά την ε, αναφορά ε, τη Σεβίλη, θυμάστε ότι ζητήθηκε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Και βέβαια, και βέβαια πρέπει να μείνει ανοιχτή. Και να ακουστούν όλε τις πλευρές. Ε, γιατί δεν κάνουμε το ίδιο και εδώ. Πριν πάρουμε την οποιαδήποτε απόφαση. Α ζητήσουμε την τοπική κυβέρνηση Ανδαλουσία και του εκπροσώπου τη επιχείρηση για να μα ενημερώσουν. Έχουμε την έκθεση που θα μα δώσει το φθινόπωρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α ακούσουμε όλε τι πλευρέ, ακούσαμε του αναφέροντε, α ακούσουμε και την άλλη πλευρά και στη συνέχεια να πάρουμε την απόφαση που είπε ο κ. Μποσινάρου ε, να μεταβούμε επί τόπου. Αλλά να ακούσουμε πρώτα όλε τι πλευρέ. Κυρία Πρόεδρε, ακολουθώντα την τακτική που φασίσαμε και στην περίπτωση τη Σεβίλη. Και εκμεταλλεύω την ευκαιρία να αναφερθώ και σε αυτά που είπαμε χθε. Ευχαριστώ. Κολέγα Κασμίρ. κύριο Κάσμαν. Ο κύριος Κάσμαν. Ε, δεν λέγαμε Κάσμιρ, Κάσμαν λέγομαι. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στι δύο λέξει. Ε, το Κασμίρ μπορεί να το φορέσει κανεί, αλλά τον Κάσμαν δεν μπορεί να το φορέσει. Άκουσα αυτή την μακροσκελή συζήτηση και θα ήθελα και εγώ να κάνω μια λογική πρόταση. Φυσικά πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά, κύριε Τουργκάη, συμφωνώ με αυτό, αλλά θα ήταν βιαστικό να επισκεφτούμε την περιοχή πριν πάει η Κομισιόν στην Ισπανία και κάνει αυτή τη διερευνητική επίσκεψη. Όταν ε, μας δώσει η Κομισιόν την έκθεσή της, θα είμαστε σε καλή θέση για να αποφασίσουμε πότε εμείς θα πάμε στην Ισπανία και τι θα κάνουμε εκεί πέρα. Γιατί συμφωνώ με τον κύριο Μάιερ ότι πρέπει να είμαστε αυστηροί αλλά επίσης δεν πρέπει να δημιουργήσουμε πανικό στον κόσμο. Ε, ε, μία ομάδα ε, ευρωβουλευτών που σπέβδουν στην ε, περιοχή αυτή για να ψάξουν δεξιά και αριστερά στέλνουν μηνύματα πανικού. Ας είμαστε αυστηροί, ας έχουμε υπομονή και ας περιμένουμε την επαληθευτική αποστολή την έκθεση της Κομισιόν για να αποφασίσουμε τότε πότε θα πάμε ε, στην Ισπανία. Αυτά λέει ο κύριος Κάσμαν. Νομίζω είναι λογικά αυτά που σας λέω. Ε, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με την ιδέα ότι θα πρέπει να επισκεφθεί μία αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στην Ουέλβα όταν κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δική της επίσκεψη. Μία ερώτηση όμως έχω να κάνω. Είναι εξαιρετική η περίπτωση. Η Κομισιόν πόσες επισκέψεις πρέπει να κάνει πριν ετοιμάσει μία πλήρη επιστημονική έκθεση. Γιατί τώρα λέει ότι θα ε, εξετάσει λέει, τα μηχανήματα με τα οποία ε, οι αρμόδιοι πηγαίνουν και μετράνε εκεί τη ραδιενέργεια και τα απόβλητα. Άλλη επίσκεψη. Νομίζω ότι το πάνελ των εμπειρογνωμόνων θα έπρεπε να εξετάσουν όλα τα θέματα τεχνικά και να καλύπτεται και το θέμα των επιπέδων ραδιενέργειας ε, ε, από αυτού. Γιατί είναι πολύ εύκολο. Με τους μετρητές Geiger μετράει κανείς τη ραδιενέργεια και μπορεί να δει σε ποιε περιοχέ η ραδιενέργεια είναι πάνω από το όριο και σε ποιε κάτω. Για να μην έχουμε τώρα κατολογίε. Και το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι η Επιτροπή Αναφορών δεν μπορεί να το παίξει διαιτητής. Ε, δεν μπορεί να πάει στην Ισπανία και να κάνει το διαιτητή μεταξύ των ε, αρχών εναντίον των κατοίκων κτλ. Για να, να παίξει αυτό το ρόλο σε άλλες χώρες. Όχι. Θα πρέπει να κρίνουμε με βάση τα γεγονότα, με τρόπο αντικειμενικό. Αν θέλουμε να είμαστε μια άξια Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάιερ. Φαντάζομαι για το θέμα της επίσκεψης, έτσι. Ναι, ναι, να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Έτσι θα ξεκινήσουμε σωστά την καινούργια θητεία. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω στο διαχωρισμό τη εξουσία και την κατανομή των αρμοδιοτήτων. Και πάντα εμεί ε, ε, δρούσαμε παράλληλα και αυτόνομα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν εδώ αποφασίσουμε ότι εμεί περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, α, αφήστε τα. Διαλύουμε την Επιτροπή και τέλειωσε υπόθεση. Δεύτερον, αυτή η συζήτηση ξεκίνησε στην προηγούμενη θητεία και συμφωνήσαμε να στείλουμε αντιπροσωπεία. Τρίτον, ο κύριος Κάσμαν πήγε στην Ισπανία με μια αντιπροσωπεία στην Βαλένθια. Και δεν πήγε έφυπος, έτσι δεν πήγε σαν υπότης. Ε, δεν ε, σκόρπισε κανένα πανικό, πήγε σε μια επίσκεψη στην Ισπανία και κατέληξε σε μια έκθεση. Άρα έτσι, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Μπορούμε να ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια, μπορούμε να επανέλθουμε στη συμφωνία που πήραμε στη συμφωνία μα σήμερα το πρωί, αλλά άλλοι είναι οι κανόνε του παιχνιδιού, δεν είναι αυτοί που είπατε. Δεν μπορεί στι 10 να συμφωνούμε το Α, στι 11 το Β. Ε, όχι, εγώ αυτό το παιχνίδι το παίζω, γιατί είμαι, νομίζω ότι είμαι σοβαρό ε, άνθρωπο. Και ε, το λέω και ενώπιον των αναφερόντων. Σήμερα το πρωί συμφωνήσαμε να εκπληρώσουμε την υπόσχεσή μα όπω εκφράστηκε στην περασμένη θητεία και να στείλουμε μια αντιπροσωπεία. Είναι αλήθεια ότι δεν την πούμε Διευρυντική Επιτροπή, θα το πούμε αντιπροσωπεία. Πάντω, εάν σε αυτή την περίπτωση πούμε δεν έχει νόημα να στείλουμε αντιπροσωπεία επιτόπου, ε, α κλείσουμε τα ρολά, α κατεβάσουμε τα ρολά. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να εκπληρώσουμε την ε, συμφωνία μα όπω ε, υπήρξε σήμερα το πρωί, όπω ελήφθη σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να δούμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να ε, ενεργήσουμε υπεύθυνα. Και κοιτάξτε για να δούμε. Εσύ ο ίδιο, Βίλη, μίλησε σήμερα το πρωί, μίλησε, συγγνώμη, ε, για διερευνητική επιτροπή. Όχι, όχι, δεν ονομάζεται διερευνητική επιτροπή. Δεν ονομάζεται επιτροπή έρευνα. Ε, πρόκειται για αντιπροσωπεία τη επιτροπή που θα επισκεφθεί μια περιοχή για να επεξεργαστεί έκθεση. Δεύτερο, το λογικό είναι το εξή. Ακούσαμε ότι όχι, δεν είμαστε, ε, ε, δεν ε, είμαστε υπόλογοι σε κάποιον, δεν ακολουθούμε κάποιον. Πάντω, αυτή τη στιγμή μια Γενική Διεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει μια συγκεκριμένη έκθεση για ένα πράγμα αποφασιστική σημασία. Ένα πράγμα είναι να πούμε, εάν θέλουμε να πάμε στην Βέλβα με επιστημονικά στοιχεία, έτσι. Όχι γιατί εξαρτώμεθα από τη δική του γνώμη, αλλά για να ελέγξουμε αυτά που θα μα πούνε, να τα δούμε επί τόπου. Και αν θέλουμε πραγματικά να επιληφθεί το πρόβλημα ή θέλουμε αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε ακριβώς και μόνο ε, εντυπώσεις. Ε, νομίζω ότι πρέπει να δράσουμε με ευθύνη, με αίσθημα ευθύνης. Εμείς δεν λέμε να μην πάμε δεν ε, ε ξαναγυρίζουμε ε, και επανερχόμαστε στην απόφαση των συντονιστών. Απλά και μόνο αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να πάμε στην Βουέλβα γνωρίζοντα και έχοντα τη διάθεσή μα ώστε να τον περισσότερα στοιχεία. Και εδώ θα έχουμε δύο εκθέσει. Μία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αξιολογίζει ε, τι αυτό που είπαν οι αρχέ και που θα ε, μα δώσει αυτή την αξιολόγηση μέσα σε λίγε εβδομάδε ή μήνε και τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που επίση μέσα σε, λίγους, σε λίγε εβδομάδε ή μήνε θα μα δώσει την έκθεση. Ε, τι λέμε, ότι η επίσκεψη αυτή να γίνει μετά, για να έχουμε και αυτά τα στοιχεία. Και αυτό είναι το λογικό και το υπεύθυνο. Αυτό είναι ο δικό μα ο ρόλος. Όχι γιατί ε, υφιστάμεθα πιέσει ή εξαρτώμεθα από την άποψη άλλων αλλά εδώ μιλάμε για, συγκεκριμένα κατευθύνσεις που θέλουν να μα οδηγήσουν τομεί, που είναι γνωστοί σε όλους θα ήθελα να πω ότι η περίπτωση αυτή αναβάλλεται συνεχώς και τώρα επιτέλους πρέπει να πάμε. Έχουμε συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες και δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό αυτό που κάνουμε. Ήδη κατά την προηγούμενη θητεία αποφασίσαμε να πάμε και τώρα ξανά είπαμε να πάμε. Φοβάμαι ότι κάτι άλλο συμβαίνει εδώ. Εγώ λέω να παραμείνουμε στην απόφαση που λάβουμε σήμερα το πρωί και να μεταβούμε επιτόπου. Κοιτάξτε, ήδη έχουμε αρκετές πληροφορίες. Φτάνουνε. Σας ευχαριστώ όλους, λέει Πρόεδρος. Σας υπενθυμίζω ότι οι συντονιστές πήρε απόφαση σήμερα το πρωί ότι θα κάνουμε δύο επισκέψεις. Άλλες επισκέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλες οι δικές μας επισκέψεις. Όπως ξεκαθαρίστηκε από τον κύριο Μαρτίνες Μαρτίνες, δεν μιλάμε για διερευνητικές αποστολές, αλλά μιλάμε για επισκέψεις, για να συγκεντρώσουμε περισσότερα στοιχεία, ούτω ώστε για να μπορούμε συνεχεία να συνομιλούμε και με τους εκπροσώπους της Κομισιόν με τα λόγου γνώσεως. Εμείς μέσω μιας επίσκεψης δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ούτως ή άλλως τα πορίσματα της ανάλυσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτως ή άλλως σήμερα το πρωί είπαμε ε, στους συντονιστές ότι θα διοργανώσουμε μία επίσκεψη εδώ στην Επιτροπή μας. Ζητήσαμε την άδεια από τις αρμόδιες αρχές. Άλλη δική μας επίσκεψη, επαναλαμβάνω, και άλλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να προχωρήσουμε όπως αποφασίσαμε. Κλείνει αυτό το σημείο και από το σημείο 21 πάμε στο σημείο 27. Eh, eh, su questa questione Οι συντάκτε θέλουν να απαντήσουν. Μια τεχνική πρόταση. Θα ήθελα να κάνω το εξή αίτημα. Μόλι ετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έκθεσή τη για την ΟΕΛΒΑ, θα ήθελα να μα αποσταλεί στην Επιτροπή Αναφορών πάρα αυτά και να ενημερωθούμε μέσω αυτή τη έκθεση και συνεχεία να ετοιμάσουμε το ταξίδι μα στην ΟΕΛΒΑ. Με ανεξαρτησία. Με ανεξαρτησία και με τα λόγου γνώσεως. Εμείς έχουμε και συμφέρον και ενδιαφέρον να διαβάσουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι ανεξάρτητο από τη δουλειά που θα κάνουμε εμείς στην Επιτροπή Αναφορών. Θα οργανώσουμε αυτή την επίσκεψη που αποφάσισαν οι συντονιστές. Οι συντάκτες της αναφοράς θέλουν να απαντήσουν entrambi. Però... Και οι δύο. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίως ε, θα ήθελα να απευθυνθώ ε, στους υπόλοιπους, ε, στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής σας που δεν είναι Ισπανοί. Για να σας πω ότι η Φερτιβέρια ΣΕΑ, αυτή η επιχείρηση, είναι μια εταιρεία που συνδέεται με ε, την, ε, που βρίσκεται στην οργάνωση ε, βιομηχανιών χημικών της περιοχής που και από άποψη οικονομική αλλά και από άποψη επιρροή στον τύπο και από πολιτική άποψη έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Εμείς θελήσαμε οι πολίτες της Ουέλβα να δημιουργήσουμε αυτό το κίνημα ε, για να καταγγείλουμε αυτή την οικονομική δύναμη, αυτή την ε, δύναμη του τύπου και δυστυχώς ε, που έχει μεγάλη δύναμη και σε τομείς της κυβέρνησης, να καταγγείλουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση. 1.200 εκτάρια καταλαμβάνουν 120 εκατομμύρια τόνοι φωσφογύψου εδώ και 40 χρόνια. Ε, και μας, έλεγαν ότι πρόκειται για υποπροϊόν και όχι για βιομηχανικό κατάλοιπο. Αποδείξαμε ότι πρόκειται για βιομηχανικά απόβλητα και ότι ε, τελικά ε, εφαρμόζεται η κοινοτική νομοθεσία επί του θέματος. Μας, μας δεν δέχονταν ότι υπάρχει κίνδυνος στο περιβάλλον δεν δέχονται ότι ε, το, τα όξινα αυτά ύδατα χύνονται στον ποταμό Τίντο. Δεν δέχονταν τίποτα. Κινητοποιήθηκαμε, από το 2002. Ε, συγκεντρώσαμε 25.000 ε, υπογραφές πολιτών από όλη αυτή την ιστορία ε, και από όλες αυτές τις διαφωνίες ωφελείται η ίδια η βιομηχανία, ο, ανεξά, ο, φορέας που είναι υπεύθυνο για τις ακτές και που υπάγεται στον οργανισμό, ε, στο φορέα για το περιβάλλον, διαφώνησε με αυτές τις απορρίψεις, αλλά τελικά η ε, κυβέρνηση της Ανταλουσίας παρέβλεψε τελείως την απόφαση αυτή. Γιατί, γιατί ο οργανισμό για το περιβάλλον μιλούσε για απορρίψει μέχρι 3 μέτρα. 25 μέτρα αφήνει η, ε, η κυβέρνηση τη Ανταλουσία. Υπάρχει απόφαση από 2005 να σταματήσουν οι απορρίψει. Βρισκόμαστε το 2009 και συνεχίζονται. Χθε, μάλιστα, χθε κατά σύμπτωση, δημοσιεύτηκε από το ε, Υπουργείο Περιβάλλοντο ότι τελικά θα εκτελεστεί η δικαστική απόφαση, αλλά δίνοντα προθεσμία μέχρι το 2002. Ε, το κλείσιμο του εργοστασίου Φερτιδέρια, στο οποίο αναφέρθηκε ο σύντροφο από, το, ε, από τους σοσιαλιστές ε, ε, αυτή η απόφαση έγινε όχι για περιβαλλοντικούς λόγους αλλά για λόγους που έχουν να κάνουν με την εργασία. Δεν υπάρχει πλέον αγορά που έχει σχέση με την αγορά, συγγνώμη. Δεν υπάρχει πλέον αγορά για τα φωσφορούχα. Άρα το κλείσιμο του εργοστασίου έχει να κάνει με τις δυνατότητες διάθεσης στην αγορά και όχι με το γεγονός ότι πλήττεται το περιβάλλον. Δεν ξέρω τι θα κάνει η φερτιδέρια. Τέλος πάντων το θέμα είναι ότι οι αρχές της Ισπανίας θα επιστρέψουν στο εργοστασίο εργοστάσιο αυτό να συνεχίσει τι απορρίψει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2012. Κοιτάξτε, ε, δεν, δεν πρόκειται να τι φοβήσουμε ούτε οι πολίτε ούτε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί τι γίνεται. Ε, ε η, η ολόκληρη πόλη της Γουέλβα ε, βρίσκεται σε αυτόν τον εκβιασμό σε σχέση με το γεγονό ότι ε, οι συνάδελφοι θα χάσουν τη δουλειά του. Μα δεν έχουν καμία σχέση όλα αυτά. Ε, η, η ίδια η επιχείρηση και η οργάνωση στην οποία ανήκει τη χημική βιομηχανία έχει μεγάλη δύναμη και έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Κα, απευθύνω έκκληση να σκεφτούμε με σοβαρότητα το ζήτημα. Για μένα ε, ήταν. Ε, ε, εγώ αισθάνθηκα ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονό ότι θα γίνει αυτή η επίσκεψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα παρακαλώ όμω να έρθετε κι εσεί, όσο το πιο γρήγορα, ανεξάρτητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να δείτε Μία και μόνο επιχείρηση, ένα εργοστάσιο, η Φερτιβέρεια. Τι κάνει στην περιοχή, σε έκταση ε, ίση με την επιφάνεια ε, της, ε, ε, της, πόλης και 500 μέτρα από την πόλη. Την επόμενη εβδομάδα θα προτείνουμε στην Επιτροπή της, τις ημερομηνίες για τις επισκέψεις. Διευκρινίζει το εξή. Δεν πρόκειται να γίνει καμία επιστημονική έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνει. Θα ελέγξει τη μεθοδολογία ε, που χρησιμοποιήθηκε στι διάφορε μετρήσει. Και τι θα μετρήσει. Μία μόνο πτυχή. Ε, τη ραδιενέργεια. Μα είναι πολλέ οι πτυχέ. Εδώ μιλάμε για ψευδάργυρο, αρσενικό και άλλα βαρέα μέταλλα τα οποία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με την επίσκεψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μετρά μόνο και εξετάζει μία μόνο πτυχή, τη ραδιενέργεια. Άρα έτσι κι αλλιώ η έκθεση δεν καλύπτει το ζήτημα. Τελειώνω. Υπάρχουν αντιφατικά στοιχεία για το ότι όταν γίνεται μία μελέτη ε, σε περιοχή τόσο πολιτικής και οικονομικής ισχύω, η ε, επιστήμη υφίσταται πιέσεις. Ακόμα και γαλλικά και ολλανδικά εργαστήρια που έκαναν μελέτες έδωσαν ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία. Ε, όσον αφορά ε, την κατάσταση των δεξαμενών. Ε, και με εκπλήσει ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο συνάδελφος είπε ότι η συμμόρφωση των, του νόμου μετά από τόσα χρόνια, γιατί το 86 ήρθε η, η, η Ισπανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από τόσα χρόνια να μην μιλάμε για τη συμμόρφωση με την νομοθεσία. Κοιτάξτε, Καταλαβαίνετε, εδώ μιλάμε για οικονομικά συμφέροντα. Η Ουέλβα ε, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τόπο. Το ποτάμι είναι θαυμάσιο. Γιατί λοιπόν θυσιάζεται στο βωμό τη της ε, ε, αγορά. Έχουμε λοιπόν ένα θέμα που αφορά το περιβάλλον και την υγεία και μια άλλη κοντόφθαλμη αντιμετώπιση που έχει να κάνει μόνο με το κέρδος και με τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, και χθε το διευκρινίσαμε. Δεν μπορούμε να απαντάμε τώρα στι ε, δεύτερε απαντήσει με δευτερολογίε και τριτολογίε. Mm, Υπενθυμίζω σε όλου του συναδέλφου επ' ευκαιρία ότι δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε δευτερολογίε και απαντήσει επί απαντήσεων γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Τέλο πάντων. Μετά από αυτό σα δίνω το λόγο παρόλα αυτά. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό και μόνο. Γιατί ε, διαστρέβλωσε τα λόγια μου ο κύριος Χαμεστή, ο οποίος ήταν και στην προηγούμενη θητεία. Ε, και κοιτάξτε, εγώ δεν αναφέρθηκα στα 20 χρόνια ε, που πέρασαν ε, και όπου δεν έγινε τίποτα. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Πρέπει να εγγυηθούμε το εξής, ότι η, το εργοστάσιο να πληρώσει ε, ε, αυτά για τα οποία είναι υπεύθυνοι. Γιατί ξέρετε τι μπορεί να γίνει, να φύγουν, να κλείσουν το εργοστάσιο, να ανοίξουν τα σχήρα του και να εξαφανιστούν. Ε, μετά τι θα γίνει, άμα φύγει, έφυγε. Ε, το 2012 το πολύ, μπορεί και πριν. Αλλά πριν φύγει, να αποζημιώσει του εργαζόμενου, να καθαρίσει την περιοχή, να δεσμευτεί ε, σε οικονομικό επίπεδο, να καθαρίσει την περιοχή. Και το ξαναλέω όλη η συζήτηση έδειξε ότι ευτυχώ δεν υπάρχει κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, αλλά μόνο για το περιβάλλον. Ας περάσουμε τώρα επιτέλους στο επόμενο σημείο, το σημείο 27 της σημερινής διάταξης. Αναφορά 0901-2008 από τον David Skinner, Σουηδικής Ιθαγένειας. Είναι παρόν ο αναφέροντας. Θέλει να πάρει το λόγο. Θα δώσω το λόγο στον συντάκτη της αναφοράς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως η αλλαγή του θέματος θα μας βοηθήσει όλους να χαλαρώσουμε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να διευκρινίσω το ερωτηματικό πάνω, δίπλα στο όνομά μου. Γεννήθηκα στην Αγγλία, αλλά εδώ και 10 χρόνια ζω κατοικώ στη Σουηδία και εργάζομαι, έχω μια επιχείρηση στο Γκότεμπεργκ. Ε, αυτή η αναφορά αφορά βασικά δικαιώματα τα οποία παραβιάζονται στην αγορά εργασίας της Σουηδίας. Μετά από διάφορες συγκρούσεις που είχαμε το 2006, ε, υπάρχουν ε, διακρίσεις και παραβίαση της ελευθερίας, της ελευθερίας και του, της ελευθερίας του συνεταιρίζεστε εμείς ε, σεβόμαστε την ανάγκη ύπαρξης ε, των συνδικάτων που χρειάζονται για την προστασία των εργαζομένων. Εγώ ε, εκπροσωπώ μια καταγεγραμμένη φιλανθρωπική επιχείρηση. Συνδεόμαστε με άλλες τέτοιες επιχειρήσεις μικρομεσαίες στην ομάδα που εκπροσωπούνται εδώ σήμερα το πρωί, το 2006 Διάφορε μικρέ οικογενειακές επιχειρήσει στη Σουηδία ε, μπήκαν στο στόχαστρο από τα συνδικάτα γιατί θέλαν να αναγκάσουν του εργαζόμενου να υπογράψουν τι συλλογικέ συμβάσει. Αυτό δεν το ζήτησαν ούτε οι εργοδότε, ούτε οι εργαζόμενοι. Και κανένα συνδικαλιστή από αυτού δεν ε, ήταν εργαζόμενο σε αυτέ τι επιχειρήσει. Αυτοί οι εργοδότε δεν μπορούν να υπογράψουν τι ε, συλλογικέ συμβάσει, γιατί έχουν μια βαθιά ριζωμένη χριστιανική πίστη. Η χριστιανική τους πίστη εμποδίζει αυτούς τους εργοδότες να μπουν σε άλλες, να ενταχθούν σε άλλες ε, οργανώσεις διαφορετικές από τις δικές τους. Έχουν βαθιές πεπιθήσεις, εδρεωμένες στο χρόνο και δεν μπορούν να συνάψουν συλλογική συμφωνία που να μην έχει σχέση με την ε, εκκλησία τους. Είπαν λοιπόν ε, μέσω των δικηγόρων τους ε, ότι οι δικές τους συνθήκες εργασίας, οι συνθήκες εργασίας που προσφέρουν είναι οι ίδιες ή και καλύτερες από τις υπόλοιπες. Ε, τα συνδικάτα απορρίπτουν ε, τη χριστιανική τους πίστη και προσπαθούν να, εκφοβ, να τους εκφοβήσουν, μάλιστα τους συκοφαντούν και μπλοκάρουν και τα, τις προμήθειές τους, ούτως ώστε να μην λαμβάνουν τα, τα αγαθά και τις πρώτες ύλες που έχουν ανάγκη. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα, χάνουν δουλειές και διάφορες επιχειρήσεις φοβούνται ότι θα μπουν και αυτές στο στόχαστρο. Αυτή η παρενόχληση των συνδικάτων είναι εντελώ απαράδεκτη. Στη Σουηδία, με βάση το Σύνταγμα, ε, το Συνδικάτο έχει το δικαίωμα να εξαναγκάσει τους εργοδότες να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις και ο εργοδότης δεν μπορεί καθόλου να προστατευθεί ε, από αυτή τη δράση αν η δράση αυτή είναι αδικαιολόγητη ή δυσανάλογη. Επειδή υπάρχει αυτή η δυσαναλογία στην αγορά είναι πάρα πολύ δύσκολο για, ένα, για μια επιχείρηση να αντιμετωπίσει τα συνδικάτα όταν εξαναγκάζουν τους εργοδότες ε, με διάφορες δράσεις, με μπλοκάρισμα των εγκαταστάσεων κτλ. να υπογράψουν τις ε, συλλογικές συμβάσεις. Το 1998 σε μια αιτήσια έκθεση ε, είπαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υπάρχει θέμα σεβασμού των δικαιωμάτων και μαζί με την Δανία και τη Γαλλία κατηγορήσαμε ότι σε αυτές τις χώρες υπάρχει παραβίαση του δικαιώματο ελευθερίας του μη συνεταιρίζεστε. Μπορούν οι εργοδότες να μην ανήκουν πουθενά. Αγαπητοί βουλευτές, η ελευθερία του μη συνεταιρίζεσαι είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και βασική ανθρώπινη αξιοπρέπεια και σε πρόσφατη αποφάσει του δικαστηρίου το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την επιβεβαίωσε. Το να μα αρνείστε αυτή την ελευθερία, ε, τα συνδικάτα ε, μα παραβιάζουν ε, το δικαίωμα ελευθερία ε, θρησκευτικής ελευθερίας. Γι' αυτό το θέμα της αναφοράς μας αφορά ένα θέμα αρχής. Και ερχόμαστε εδώ να κάνουμε έκκληση ε, ενώπιον του Κοινοβουλίου να εξετάσει αυτό το θέμα. Η οδηγία, 09, η οδηγία του 2000 απαιτεί να μην γίνονται τέτοιου τύπου παραβιάσεις και οποιαδήποτε δράση, ε, απεργία ή οποιαδήποτε άλλη, ε, θα πρέπει να είναι δικαιολογημένη, ανάλογη κτλ. Όταν υπάρχουν παραβιάσεις της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και όταν δημιουργείται ένα ταπεινωτικό ε, και εχθρικό περιβάλλον είναι πρόβλημα. Αυτό ακριβώς συνέβη σε εργαζόμενους και εργοδότες. Και με κάθε ταπεινοφροσύνη σας προτείνουμε αυτή η σημαντική οδηγία να εφαρμοστεί, να εφαρμοστεί και για αυτή την αναφορά. Μπορεί κάποιος να μας ρωτήσει γιατί δεν προσφεύγεται στα σουηδικά δικαστήρια. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν νομίζω ότι σε ένα σουηδικό δικαστήριο θα μας αντιμετωπίσουν με βίκο νους. Γιατί το εργατικό δίκαιο ε, στη Σουηδία είναι άδικο σε τέτοιου τύπου διαφορές. και τα συνδικάτα απλώς ε, ασκούν τα δικαιώματα που τους έχουν δοθεί δια νόμου. Αντίθετα αυτή η ελευθερία του μη συνεταιρίζεστε μας αρνείται. Μας την αρνούνται. τα συνδικάτα έχουν ε, δικαίωμα ε, εξασφαλισμένο μέσω του συντάγματος. Επομένως, δεν έχει κανένα νόημα εμείς να προσφύγουμε σε δικηγόρο και να πάμε σε δικαστήριο. Χρειάζονται κάποιες αλλαγές ε, στην σημερινή Σουηδική εργατική νομοθεσία, ούτως ώστε να δοθεί σε αυτούς τους εργοδότες μια κάποια προστασία εναντίον αυτής της διάκρισης και της παρενόχλησης. Αγαπητοί βουλευτές, κυρία Πρόεδρε, σας ζητούμε η Επιτροπή να γράψει μια επιστολή στην κυβέρνηση και να καταδείξει ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Οδηγία θα πρέπει, που θα έπρεπε να είχε γίνει σεβαστή από όλα τα κράτη-μέλη μέχρι το 2003 να εφαρμοστεί και στη Σουηδία και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία της Σουηδίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Σίγουρα η Επιτροπή Αναφορών θα έρθει σε επαφή με τις Σουηδικές Αρχές. Η Κομισιόν είναι εδώ παρούσα. Θα ήθελα ο εκπρόσωπός της, δεν τολμώ να πω το όνομά του, γιατί θα το προφέρω λάθος, ε, θα ήθελα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν να πάρει το λόγο. Είναι παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, το όνομα μου είναι Στέφανο και ο κύριος Φένστρα που αναφέρεται εσείς κάθε δεξιά μου. Ε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον ε, Τούντα για την ε, παρουσίαση αυτής της υπόθεσης. Εμείς το θέμα αυτό το πήραμε πάρα πολύ σοβαρά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί πράγματι άπτεται αρκετών τομέων. Είχαμε αρκετές διαβουλεύσεις ε, με τους συναδέλφους μας. Το θέμα των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι ένα θέμα που διατρέχει πολλές γενικές διευθύνσεις. Η ίδια η αναφορά νομίζω ότι είναι σαφέστερη. Ακούσαμε από τον αναφέροντα το θέμα της ε, των θρησκευτικών διακρίσεων. Μας το εξήγησε αυτό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη δική μας την απάντηση, όπως ε, είπε και ο ίδιος, κάνουμε αναφορά στην οδηγία 2078 στα δικαιώματα των εργοδοτών. Και δεν θέλουμε να ε, αποκλείσουμε ότι αυτή υπερισχύει και των ε, θεμάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει λοιπόν να επανέλθω στην ε, νομική μας υπηρεσία, η 2078 η οδηγία αυτή κατ' ουσίαν αφορά τη συμμετοχή ή την ε, εμπλοκή σε ενώσεις. Associations. Αλλά για μας δεν είναι σαφές κατά πόσον εδώ πρόκειται για ε, σχέσεις συλλογικών συμβάσεων. Κατά πόσον, δηλαδή εταιρείε οι οποίες συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις κατά πόσον καλύπτονται από αυτήν την οδηγία ή όχι. Αυτά λοιπόν ε, τα θέματα που έθιξε ο αναφέρον θα τα εξετάσουμε, αλλά εγώ προσωπικά θέλω να σας πω ότι έχω αμφιβολίες για το κατά πόσο στην περίπτωση αυτή ισχύει αυτή η οδηγία. Κατόπιν, πέρα από την οδηγία, αν δούμε και άλλα θέματα, υπάρχει το θέμα των ε, συλλογικών διαπραγματεύσεων του ε, δικαιώματος ε, του, της ελευθερίας του μη συνεταιρίζεστε, στην οποία αναφέρθηκε ο αναφέρον. Βεβαίως ε, και όλα αυτά εμπίπτουν στο θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Κομισιόν δεν μπορεί να παρέμβει αν δεν πρόκειται σαφώς για ένα θέμα που έχει σχέση με το κοινοτικό δίκαιο. Από νομικής λοιπόν πλευράς η οδηγία είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις κατά πόσον το θέμα αυτό εμπίπτει στην εμβέλεια της οδηγίας ή όχι. Ίσως θα έπρεπε ο αναφέρον να μας γράψει περισσότερα στοιχεία για το θρησκευτικό στοιχείο του θέματος και θα το εξετάσουμε. Βεβαίω ε, έκανε ο αναφέρον ε, παρατηρήσεις για το κατά πόσον έχει νόημα να απευθυνθούν σε Σουηδικό Δικαστήριο όχι. Πάνω σε εγώ θέλω να πω ότι φυσιολογικό θα ήταν να καταφύγουν στα Σουηδικά Δικαστήρια και εάν δεν ικανοποιηθούν να ζητήσουν παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όπως είπε όμως και ο αναφέρον, επειδή το θέμα αυτό εξετάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, είναι πολύ πιθανόν να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο ε, επαναλαμβάνω, αυτό είναι ένα φυσιολογικό δρόμο για μια τέτοια είδου περίπτωση. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, αλλά αν θέλετε, πολύ ευχαρίστω είμαι στη διάθεσή σα για να απαντήσω σε ερωτήσει. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας παρακαλώ δεν θα θέλατε πρώτα να μιλήσουν όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές ε, και ενδεχομένω ξανά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλο να απαντήσετε εσείς, κύριε Συντάκτη. Θα είμαι πολύ σύντομη. Κοιτάξτε, πράγματι θα πρέπει να κάνουμε αυτό ε, που μας συμβουλέψετε να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, αλλά εγώ διαμαρτύρομαι. Εδώ γίνεται χρήση της ε, χριστιανικής ε, πίστης για να τεκμηριώσει μια υπόθεση. Στη Δανία εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τον συνδικαλισμό. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ δυσάρεστο το να επικαλείστε την ε, χριστιανική πίστη ε, ως επιχείρημα για να στηρίξετε την ελευθερία του μη συνεταιρίζεστε. Και ε, θα ήθελα παρακαλώ αυτό να γραφτεί στα πρακτικά, γιατί εδώ πραγματικά γίνεται κατάχρηση ε, της χριστιανικής πίστης και αυτό είναι λάθος, θεωρώ ότι όλοι μας εδώ ε, είμαστε χριστιανοί. Ο κύριος Λούντβινγκσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ για να σας δώσω τη γνώμη μου. Η εργατική νομοθεσία της Σουηδίας βασίζεται σε αποφάσεις του Σουηδικού Κοινοβουλίου, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι διαπραγματεύσεις των συλλογικών συμβάσεων ε, υποστηρίζονται από το Σουηδικό Δίκαιο. Και από ό,τι βλέπω οι συντάκτες της αναφοράς δεν υπόκεινται σε διακρίσεις. Τα συνδικάτα της Σουηδίας σε καμία περίπτωση δεν εξαναγκάζουν τον κόσμο να γίνουν μέλη αλλά ως ένας από τους ε, κοινωνικούς εταίρους, τα συνδικάτα προσπαθούν απλώς να προασπίσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τα συνδικάτα έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν ε, σε δράση εναντίον των ε, επιχειρήσεων που αρνούνται να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις. Αυτή η δράση δεν αφορά ποτέ συγκεκριμένα άτομα, ιδιώτες. Και ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος μπορεί να, να καταλάβει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Επιτροπή ας πούμε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή την Επιτροπή Αναφορών για να εξαιρεθούν αυτές οι επιχειρήσεις από τις επιταγές του νόμου, της εργατικής νομοθεσίας. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Κοιτάξτε εδώ, πρόκειται για μια πολύ περίεργη και ειδική αναφορά. Ως σοσιαλιστής γνωρίζω ότι η νομοθεσία στη Σουηδία είναι από τις ε, πλέον προχωρημένες, από τις καλύτερες. Οι σχέσεις ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία ακολουθούν ένα συγκεκριμένο δρόμο και αυτό ε, προσέδωσε στη χώρα πλούτο, πολιτισμό, παιδεία και εμείς απ' έξω ζηλεύουμε την εξέλιξη της Σουηδίας. Τώρα, ε, το να ε, γίνεται χρήση της Εκκλησίας ως στοιχείο, αυτό νομίζω ότι είναι λάθος, γιατί κατά τη δική μου τη γνώμη, ε, όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις, είναι παντελώς αδιάφορο κατά πόσον ο εργαζόμενος έχει θρησκευτική πίστη ή σχέση με την Εκκλησία ή όχι. Η προάσπιση των δικαιωμάτων του δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκευτική πίστη. Εγώ τη γνωρίζω τη Σουηδία, τη θαυμάζω και οι σχέσεις εργοδοτών εργαζομένων στη Σουηδία είναι πρότυπο για πολλές χώρες της Ευρώπης. Γιατί πραγματικά είναι πολύ καλές οι σχέσεις. Παραδείγματος χάρη αν ε, κάποιος ε, απολυθεί, αυτό δεν θεωρείται, δεν εκλαμβάνεται ως ε, ότι συνέβη κάτι επειδή ήταν δούλος. Ε, γι' αυτό λοιπόν εγώ πραγματικά μας πω ότι έχω πολλές επιφυλάξεις όσον αφορά αυτή την αναφορά. Ε, ο, οι, εργο, εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις ε, επιλέγονται με βάση το θρησκευτικό τους, ε, ε, το, τις θρησκευτικές αντιλήψεις τους ή όχι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η απάντησή σας, η απάντηση στην ερώτησή σας είναι όχι. Σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζεται, δεν επηρεαζόμαστε από κάτι τέτοιο. Ε, εγώ έχω και Ρουμάνους μάλιστα εργαζομένους. Ε, είμαστε μία χαρούμενη οικογένεια στην επιχείρηση. Ε, αντιμετωπίζουμε όλο τον κόσμο με δικαιοσύνη ε, και δεν υπάρχουν ε, συνδικαλιστές καθόλου σε αυτούς. Για να απαντήσω και στην κυρία Άλκιν, η οποία λέει τι σχέση έχει η χριστιανική πίστη με αυτό. Να μην ξεχνάτε ότι στη χάρτα ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάρχει και το δικαίωμα της αντίρρησης. Αυτό το δικαίωμα θα πρέπει να, σεβαστεί, να γίνει σεβαστό είναι εναντία στη συνείδησή μου ω εργοδότη. Γιατί έχω τα συνδικάτα που μου λένε πρέπει ντε και καλά να υπογράψω αυτέ τι συλλογικέ συμβάσει. Εγώ λέω, συγγνώμη. Ε, εγώ ανήκω στην ε, εκκλησία Τάδε, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να υπογράψω αυτέ τι συλλογικέ συμβάσεις. Έχω την πίστη μου. Και με μπλοκάρουν. Αλλά εγώ έχω το νομικό δικαίωμα να μην κάνω κάτι τέτοιο. Ο νόμος όμως με αφήνει έκθετο. Δεν μπορώ να αντιταχθώ στην ε, στάση αυτή των ε, συνδικάτων. Ε, είναι απίστευτο αυτό το δικαίωμα που έχουν δια συντάγματος, δια νόμου τα συνδικάτα. Είναι απίστευτο που συμβαίνει αυτό στη Σουηδία, αλλά συμβαίνει. Η Σουηδία προσπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και παντού στον κόσμο παίζει αυτό το ρόλο, σηκώνει αυτό το δαυλό. Χαίρομαι πάρα πολύ, αλλά είναι θέμα χριστιανική πίστη αυτό και θα πρέπει να γίνει σεβαστή η χριστιανική πίστη. Ο Υπουργό Εργασία θέλει να μα βοηθήσει. Κατανοεί τα, επιχειρη... τα επιχειρήματά μα. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν δεν αλλάξει, αν δεν τροποποιηθεί η εθνική νομοθεσία. Να υπάρχει δηλαδή μια ενδιάμεση διάταξη ε, ούτω ώστε να μπορούν ε, εργαζόμενοι και εργοδότες να εκφύγουν και να τεθούν εκτός μιας συλλογικής σύμβασης. Στο άρθρο 1, θα ήθελα να σας πω κύριε, ε, της οδηγίας αυτής λέγεται ότι υπάρχει γενικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της ε, διάκρισης λόγω ε, θρησκείας ή πίστης. Ε, αυτό το λέει το άρθρο 1 αυτής της οδηγίας του 2000. αν υπάρχει διάκριση νομίζω ότι πρέπει να γίνει σεβαστή αυτή η οδηγία γιατί αυτή η οδηγία μιλάει για τις διακρίσεις. Πρόεδρος. Το θέμα αυτό δεν αφορά τη θρησκεία. Γιατί αν αφορά τη θρησκεία, εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι και η αναφορά σας δεν θα ήταν παραδεκτή. Νομίζω ότι το βασικό σας επιχείρημα είναι πολύ, κάτι πολύ πιο ευαίσθητο, κάτι πολύ πιο λεπτό και μπορούμε να το εξετάσουμε. Δηλαδή ότι παραβιάζεται από ένα κράτος μέλος, α, παραβιάζονται συνθήκες και αρχές ε, που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς, παραβιάζεται η ελευθερία του, του συνεταιρίζεστε και το συνεπακόλουθό της που είναι η ελευθερία του μη συνεταιρίζεστε και η θρησκευτική ελευθερία. Επομένως, μέσα από τις ε, έρευνες και διερευνητικές αποστολές που κάνουμε εμείς, εμείς στην Επιτροπή θα εξετάσουμε αν το σουηδικό σύστημα παραβιάζει αυτές τις βασικές αρχές. Ανεξάρτητα από τους λόγους. Έτσι. Μας ε, υποβλήθηκε και ένα σημείωμα ε, για αυτό το θέμα. Εξού και η ερώτηση της κυρίας Παλιαδέλη. Στο το σημείωμα αυτό αναφέρεται η νομοθεσία η Σουηδική στον αρμόδιο τομέα. Και εκεί γίνεται λόγος για την υποχρέωση ε, εγγραφής σε κάποιο συνδικάτο. Ε, αυτό μας ενδιαφέρει. Τώρα το θέμα του αν έχει κάποιος πίστη ή όχι, αυτό είναι κάτι άσχετο. Δεν μας ενδιαφέρει. Επομένως το σημείο αυτό παραμένει ανοιχτό. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Πάμε στο επόμενο σημείο, που είναι το σημείο 28 της ημέσιας διάταξης. Ο αναφέρον είναι παρόν, έτσι δεν είναι. Ο κ. Κίνγκ. Δίνω το λόγο στον κ. Κίνγκ. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τη δική μου την ε, αναφορά, είναι ξεκάθαρο το ποιο είναι καταρχήν το θέμα. Εδώ δεν πρόκειται για μία περίπτωση ότι υπάρχει αμφιβολία για το κατά πόσον υπήρξε παραβίαση ή όχι. Okay. Λοιπόν, ε, εδώ είναι μια περίπτωση όπου η Κομισιόν έχει δεχθεί επανειλημμένα ότι υπάρχει παραβίαση και η Κομισιόν κάνει ό,τι μπορεί ε, για να ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση. Στις 5 Μαΐου του 2007 η Κομισιόν συμφώνησε ότι το, η νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο παραβιάζει την ε, κοινοτική νομοθεσία και εκεί αναφέρεται ότι οι σύζυγοι ε, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να ε, μπουν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ε, βίζα. Όμως το δίκαιο της Αγγλίας δεν δέχεται κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν το 2008 η Κομισιόν ενέκρινε μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας αυτής του 2000, της 2004 38 και παράγραφος η σχετική επαναλαμβάνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραβιάζει το 5.2 ε, του κανονισμού εδώ ε, είναι δυσάρεστο το ότι παρότι διαπιστώθηκε επανειλημμένο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ε, παραβιάζει το δίκαιο, ε, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα διαδικασία επί παραβάση. Και μάλιστα η Κομισιόν συνεχίζει να βρίσκει κάποιε προφάσεις για να μην δρομολογήσει αυτή τη διαδικασία. Πρόσφατα η Κομισιόν με επιστολή ανακοίνωσε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εξετάσει κάποιε τροποποιήσει στην κείμενη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου που εγκρίθηκε πρόσφατα έτσι λοιπόν είναι σαφές, ακόμα και αν δει κανείς επιπόλαιο το όλο θέμα, ότι έχουν άμεση σχέση ε, με την ε, νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, γιατί υπήρξαν κάποιες τροποποιήσεις, όχι όμως σε αυτό το θέμα. Η Κομισιόν το να ισχυρίζεται ότι χρειάζεται χρόνο για να εξετάσει αυτά τα θέματα είναι απλά ε, Και η δική μου η αναφορά εκρεμεί εδώ και τρία χρόνια, ενώ ο χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει κανείς στο δικαστήριο είναι λιγότερος από δύο χρόνια. Είναι λοιπόν εντελώ απαράδεκτο το να καθυστερεί τόσο πολύ διαδικασία επί παραβάση, ενώ δεν χρειάζεται ανάλυση άλλων ε, δευτερευόντων ε, θεμάτων. Και θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Επιτροπή ε, να ε, τοποθετηθεί για το χρόνο που χρειάστηκε η Κομισιόν και να καλέσει την Κομισιόν να κάνει το πρώτο βήμα στη διαδικασία επιπαραβάση, δηλαδή ε, να στείλει η ε, Κομισιόν επίσημη επιστολή πάρα αυτά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και θα ήθελε το θέμα αυτό μετά από έξι μήνε να ξαναμπεί στη μέση διάταξη για να ελέγξουμε το μεταξύ τι είδου πρόοδο έχει επιτευχθεί στι δράσει τη Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν απαντήσω στα όσα είπε ο κύριος Κίνγκ, θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η συγκεκριμένη αναφορά που έχει προσαρτηθεί σε ένα φάκελο άλλων 6-7 αναφορών ε, αφορά ε, μία σειρά από καθυστερήσεις. Θα μιλήσω καταρχάς για τις θεωρήσεις, αλλά εν συνεχεία θα μιλήσω για τις ε, καθυστερήσεις. Είναι σωστό αυτό που είπε ο κύριο Κίνγκ, ότι η Κομισιόν κατά, κατά επανάληψη της, του είπε ότι υπάρχει παραβίαση στην Βρετανική νομοθεσία ε, που ε, μετέφερε την Οδηγία 2004-38 για την ε, κίνηση των ε, μελών της οικογένειας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια νέα οδηγία που κωδικοποίησε το σώμα του κοινοτικού κεκτημένου σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα και αντικατέστασε, αντικατέστησε διάφορες πράξεις του κοινοτικού δικαίου. Αυτή η οδηγία υιοθετήθηκε το 2004 και έπρεπε να εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του Απριλίου 2006. Όλα τα κράτη-μέλη δεν, έχουν, ε, δεν εφάρμοσαν ε, εγκαίρως ε, της, αυτή την νομοθεσία. Ε, ξεκινήσαμε διαδικασίες επί παραβάση τελευταία διαδικασία έκλεισε το, ξεκίνησε, έκλεισε μάλλον τον Νοέμβριο του 2006. Η Κομισιόν υιοθέτησε και μία έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας ε, που εντόπισε περίπου 11.000 παραβάσεις στα κράτη-μέλη. 11.000. Η παράβαση του κυρίου, που υπέστη ο κύριος Κίνγκ είναι μία από αυτές τις 11.000. Πρέπει να προσεγγίσουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε 11.000 διαδικασίε επί παραβάση. Επομένω, λάβαμε την απόφαση να συγχωνεύσουμε όλε αυτέ τι παραβάσει, ε, να, λοιπόν, ε, να στείλουμε μία επίσημη επιστολή ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλη μία επιστολή στο άλλο, στα άλλα κράτη-μέλη, αντί για 11.000 επιστολές. Στην έκθεση αυτή του Δεκεμβρίου η Κομισιόν είπε ότι υπάρχουν προβλήματα με τις θεωρήσεις ε, και αυτά είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα ε, παράβασης ε, των δικαιωμάτων των μελών της οικογένειας των Ευρωπαίων πολιτών. Και πώς αντιμετωπίσαμε το θέμα στις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της οδηγίας. Μπορείτε να τις βρείτε όλοι οι βουλευτές της Επιτροπής Αναφορών. Με αυτόν τον τρόπο ε, προσπαθούμε να δώσουμε οδηγίες ε, ούτω ώστε να μην συμβαίνουν αυτά τα προβλήματα. Οι τροπολογίες της ε, Βρετανικής νομοθεσίας που έγιναν εφαρμοστές τον Ιούνιο του 2009 δεν αφορούν άμεσα το τμήμα της Βρετανικής νομοθεσίας που αφορά την εξαίρεση των θεωρήσεων αλλά εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε όλα τα θέματα παράλληλα, όλα τα προβλήματα των παραβάσεων παράλληλα. Δυστυχώς βεβαίως για τον κύριο Κιν, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις ε, σε ό,τι αφορά την πρόοδο ε, για το δικό του θέμα. Αυτά έχω να πω για τη συγκεκριμένη αναφορά. Κυρία Γουόλης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, εγώ ε, δεν είχα πρόθεση να ασχοληθώ με αυτή την αναφορά, αλλά από ό,τι άκουσα, εδώ πρόκειται για έναν υπήκο του Ηνωμένου Βασιλείου. Και είναι ένα θέμα για το οποίο παίρνω πάρα πολλέ επιστολέ από ψηφοφόρου τη εκλογική μου περιφέρεια. Χαίρομαι με αυτά που είπε η Κομισιόν και άκουσα ότι θα υπάρξει ε, συγχώνευση όλων των ε, διαμαρτυριών και των αναφορών για να ε, δρομολογηθεί η διαδικασία επί παραβάση. Εγώ όμως θα ήθελα πολύ να μάθω πότε θα γίνει αυτό. Πότε θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Δεν βλέπω να υπάρχει κανείς το... Okay. Κοιτάξτε, η Επιτροπή με την πεπατημένη ε, έρχεται σε επαφή με τα κρατημέλη για να τους ανακοινώσει όλες ε, τις ε, παραβιάσεις. Την πρώτη συνάντηση την έχουμε την επόμενη εβδομάδα και η επιστολή προς το Ηνωμένο Βασίλειο όπου αναφέρονται όλα τα θέματα παραβιάσεων. Αυτή η επιστολή υπολογίζουμε ότι θα σταλεί γύρω στις 4 με 6 εβδομάδες. Είπατε... ότι θα γίνει μια συνάντηση με τα κράτη-μέλη. Υπάρχει περίπτωση να μην σταλεί επιστολή ανάλογα με τι θα συμβεί στην επίσκεψη, στην συνάντηση με τα κράτη-μέλη. Τι συμβαίνει λοιπόν, τι θα συμβεί. Θα στείλουμε επιστολές σε όλα τα κράτη-μέλη που οι επιστολές αυτές θα αφορούν και τις 11.000 περίπου παραβάσεις και θα ζητήσουμε σχόλια και παρατηρήσεις. Γιατί τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν και με βάση τις ε, παρατηρήσεις τους και την τεκμηρίωση που θα μας στείλουν, τις διευθυνήσεις που θα μας ε, δώσουν, μπορεί να μειωθεί ο κατάλογος των παραβάσεων. Αλλά όταν υπάρχει α, πράγματι παράβαση του κοινοτικού δικαίου, ε, αυτή η συγκεκριμένη παράβαση θα καλύπτεται από προειδοποιητικές επιστολές. Επομένως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι παραμένει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Πάμε τώρα στα σημεία 29 έως 32 πρέπει να τα διεκπαιρεώσουμε. Γιατί αφορούν την αρμοδιότητα της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να τα διεκπαιρεώσουμε γρήγορα για να περάσουμε στι επόμενες που είναι παρόντες και οι συντάκτες. Πάμε λοιπόν πάρα αυτά στην 29. Ο κύριος Μεντούνα. Okay, basically... Θα καλύψω λοιπόν όλα τα ζητήματα αυτά, είτε περισσότερα από τα ζητήματα, σε μία παρέμβαση. Πρώτα, να σας πω ότι και εμείς και εσείς παίρνετε πολλές διαμαρτυρίες όσον αφορά τις καθυστερήσεις ε, για τις αιτήσει ε, για τη διαμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφέστατη. Υπάρχουν αυστηρές προθεσμίες στην κοινωτική νομοθεσία. Μέσα σε 6 μήνες από τους, ε, στους τρίτους και τις οικογένειές τους, ενώ οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ίδια μέρα. Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από αρκετό καιρό αποφάσισαν να μεταφέρουν ορισμένους αρμόδιους υπαλλήλους από το τμήμα που ασχολείται με, τις, ε, με το θέμα αυτό ε, και να τους μεταθέσουν σε μια άλλη υπηρεσία. Αυτό οδήγησε τρομερές καθυστερήσεις. Άρα είχαμε καθυστέρηση πάνω από ένα έτος και αυτό σε συστηματική βάση. Και αφορούσε, αυτή η κατάσταση αφορούσε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που υπέβαλαν τις αιτήσει. Η Επιστροπή παρενέβη προς τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Ζητήσαμε να μας δώσουν να λάβουν υπόψη ε, τις διατάξεις πάσης φύσεως έτσι ώστε να συμμορφωθούν με την κατάσταση ε, αυτή, ε, να ξεκαθαρίσουν με τις καθυστερήσεις να πιο γρήγορα και στην ουσία να ε, εφαρμόσουν σωστά την οδηγία 38 του 2004 καθώς επίσης να μας δώσουν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Αυτό έγινε το Μάρτιο, οι αρχές του Ηνωμένου Βασίλειου απάντησαν το Μάιο δέχτηκαν ότι υπήρξαν αυτές τις καθυστερήσεις όσον αφορά την χορήγηση της άδειας διαμονής, αναγνώρισαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, εφάρμοσαν ένα συνολικό σχέδιο με, με στόχο να συμμορφωθούν με την κοινωτική νομοθεσία μας το Δεκέμβριο 2009, ε, ε, ε, αύξησαν σημαντικά τον αριθμό των υπαλλήλων που θα ε, διεκπαιρεώνουν τις υποθέσεις αυτές η αύξηση λοιπόν των πόρων σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη κατάρτιση η ε, ε, επεξεργασία ε, των υποθέσεων αυτών έχει ήδη οδηγήσει σε, σε επιτυχή αποτελέσματα και από τις 500 υποθέσεις την εβδομάδα το Φεβρουάριο πήγαμε σε 1500 το Μάιο. Είδαμε λοιπόν ότι Ηνωμένες, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι αρχέ του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν αναλάβει τη δέσμευση να προχωρήσουν σε αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματο. Και όμως από την άλλη πλευρά ε, παίρνουμε μηνύματα που δείχνουν ότι αρχίζουν να δίνονται ε, αιτήσει πιο γρήγορα. Ε, Άδειε. 1500 ε, επίσημες προσφυγές πήραμε επίσημες καταγγελίες. Όλο αυτό ε, δείχνει τη σοβαρότητα του προβλήματος και ε, ε, αναγνωρίζουμε τη σοβαρότητα. Το πιο σημαντικό είναι ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει κανείς τα ταχυδρομικά την αίτησή του και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να επισυνάψει. Στέλνει λοιπόν στο Υπουργείο Ιστορικών με το ταχυδρομείο ο ετών. Δυστυχώς όμως ε, για τους ετούντες μέρος της αίτηση, ε, μέρος των εγγράφων ε, πρέπει να είναι το επίσημο διαβατήριο, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις βρέθηκε στο γραφείο υπαλλήλων στο Λίβερπουλ για πάνω από ένα χρόνο. Καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο πρόβλημα. Και γι' αυτό οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου εισήγαγαν από τον Ιούνιο του 2009 ε, μία, έδωσαν δηλαδή μία συγκεκριμένη διεύθυνση email όπου οι ετούντες θα ζητούν την επιστροφή του διαβατηρίου τους μέσα σε 10 χρόνια. Άρα, άλλαξαν τη διαδικασία, δεν κρατούν πλέον το πρωτότυπο ε, όσο εξετάζεται η υπόθεση. Και όπως σας είπα, ε, έχουν προβλέψει και μια ηλεκτρονική διεύθυνση, αλλά και μια συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή, την οποία παίρνει κανείς τηλέφωνο, παίρνει το τηλέφωνο αυτό και ζητά το διαβατήριό του. Θέλω να σα πω γενικέ γραμμέ ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τα μέτρα τα οποία έλαβαν οι αρχέ του Ηνωμένου Βασιλείου για την αντιμετώπιση του προβλήματο. Ε, θα εξακολουθήσουμε ε, να παρακολουθούμε την εφαρμογή όλων αυτών ε, στην πράξη ε, και εξακολουθούμε να παίρνουμε ε, δεκάδες ε, παράπονα, αλλά όπως σας είπα, ορισμένες καταγγελίες ε, εξετάσαμε ορισμένες καταγγελίες και, φαίνεται ότι ήδη η κατάσταση έχει αρχίσει να αποκαθίσταται. Αυτό καλύπτει όλα τα ζητήματα όσον αφορά την 28. Ε, κάτι άλλο τώρα που έχει να, που έχει ε, να κάνει με την ενσωμάτωση του Εθνικού Δίκαιου του Ηνωμένου Βασιλείου τη Οδηγία 38-2004, που έχει να κάνει με την 29 και με την ε, μόνιμη διαμονή. Όπω τα γνωρίζετε ενδεχομένω, η οδηγία για πρώτη φορά ε, εισάγει ένα γενικό δικαίωμα μόνιμη άδεια παραμονή για αυτού που ζουν το συγκεκριμένο κράτο, πάνω, ε, μέλος, κράτος πάνω από πέντε χρόνια. Το Ηνωμένο Βασίλειο ερμήνευε, η ερμηνεία μάλλον που δίνει το Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτή τη συγκεκριμένη διάταξη της οδηγίας, ε, στην ουσία αποκλεί όλους τους πολίτες από τα νέα κράτη-μέλη από αυτό το δικαίωμα. μέχρι το 2009 για τις, όλες τις χώρες πλήν της Βουλγαρίας και Ρουμανίας και εκεί πήγαινε στο 2012. Δηλαδή, ερμηνεύει ότι τα, ε, ερμηνεύει την διάταξη αυτή ότι, ότι τα άτομα αυτά πρέπει να μένουν ε, ω πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για πέντε χρόνια. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για το τέλο ε, του πενταετού διαστήματο. Τότε πρέπει να είναι, ε, να ανήκουν, να είναι υπήκοοι ενό κράτου μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι όλο το διάστημα ε, των πέντε ετών. Και στο παρελθόν ήρθαμε σε επαφή με, τον, με τι αρχέ του Ηνωμένου Βασιλείου. Του επιστήμονε προσοχή σε αυτή τη διαφορά ερμηνεία διαφώνησαν με τη δική μα ερμηνεία και αυτό ήταν ένα ζήτημα το οποίο καλύφθηκε και, καλύφθηκε και στην έκθεση ως, όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας και ε, ε, αυτό το σημείο λοιπόν ε, θα καλυφθεί σαφώς και στη διαδικασία παράβασης που θα κινηθεί κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Γιατί ήδη ήρθαμε σε προηγούμενες επαφές, σε εκ των προτέρων επαφές με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και έχουν γίνει ξεκάθαρες οι θέσεις. Σταματήστε με, διακόψτε με, λέει ο εκπρόσωπο εάν ε, ε, έχω ξεπεράσει τα όρια, τα χρονικά όρια. Λοιπόν, Τώρα άλλο, ένα άλλο ζήτημα αφορά ε, το 31 για τα μέλη οικογένειας ε, ανθρώπων που έχουν άδεια διαμονής και κατά πόσον ε, είναι, είναι η, αναφορά του κυρίου Κίνγκ ε, και κατά πόσο απαλλάσσονται από την ε, υποχρέωση θεώρησης. Αυτά που είπα λοιπόν στην 31. Uh, Όσον αφορά την 32. Εδώ έχουμε και θέματα που αφορούν την αίτηση, την αναφορά του κυρίου Κίνγκ και την 31. Και εδώ έχουμε να κάνουμε το ευρύτερο θέμα ε, της πολιτικής θεωρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά δηλαδή, τη θεώρηση εισόδου όπου ε, φαίνεται ότι ε, η καταγγελία αφορά το γεγονό ότι δεν διευκολύνουν καθόλου τη διαδικασία οι εθνικέ αρχέ. Έχουμε πάρει πάρα πολλέ ε, καταγγελίε για το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα το οποίο εξετάστηκε και στην έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας το Δεκέμβριο 2008, αλλά και στις κατευθυντήριες γραμμές του Ιουλίου του 2009. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτά τα δύο έγγραφα από κοινού με ε, την σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη συνεργασία ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα κράτη-μέλη, θα μα βοηθήσει να δούμε και τα δύο αυτά ζητήματα. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι το ζήτημα αυτό θα, συζητηθεί με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και θα συμπεριληφθεί ε, στην επίσημη προειδοποιητική αποστολή. Επιστολή. Αλλά αν τώρα στο μεταξύ οι αρχέ του Ηνωμένου Βασιλείου συνειδητοποιήσουν το πρόβλημα και προχωρήσουν τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων, τότε τα πάντα θα έχουν λυθεί. Ε, εδώ ε, αυτές είναι οι αναφορές τι οποίες ευσταθούν τα επιχειρήματα των αναφερόντων. Κυρία Γουόλης, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προσπάθειά σας ε, να ασκήσετε πίεση στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Προφανώς είχατε μια κάποια επιτυχία ε, όσον αφορά την πρόοδο σε ορισμένου τομεί. Δύο ερωτήσει θέλω να έχω που θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε. Πρώτα απ' όλα, το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, έχω δίκιο να θεωρήσω ότι είναι ε, το μόνο κράτο μέλο το οποίο ζητάει τα πρωτότυπα διαβατηρίων τα οποία υποστέλλονται με το χειδρομείο, στερώντα με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα μετακίνηση ε, των ε, πολιτών. Και δεύτερο, για να καταλάβω τι γίνεται όσον αφορά την ερμηνεία αυτού του πενταετού χρονικού διαστήματο. Δηλαδή να έχει μείνει κανεί πέντε χρόνια ω ε, υπήκο κράτου μέλου. Αυτό το ζήτημα πρέπει να αποφασιστεί σε, νομική, σε νομικό επίπεδο. Εδώ δεν έχω καταλάβει. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία παράβαση. Και τι ακριβώ συμβαίνει. Θα σα ήμουν ευγνώμων να μπορούσατε να το ξεκαθαρίσετε το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ την κυρία Γουόλης. Για να διευκρινίσω και τα δικά μου ερωτηματικά, αλλά και τα ερωτηματικά των συναδέλφων. Με την παρέμβαση που ακούσαμε από τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης, διεκπαιρεώσαμε όλες τις αναφορές μέχρι την υπαριθμό 32, γιατί το θέμα είναι το ίδιο. Οι παραβιάσεις των οδηγιών 2004 ε, κάθετος 38. Ε, διάφορες παραβιάσεις διαφόρων κεφαλαίων. Επομένως, η Κομισιόν θα γράψει για να τις δοθούν ε, ξεκαθαρίσει από τις Βρετανικές Αρχές και θα γράψει για όλες τις αναφορές. Σωστό αυτό? Όχι. Όχι. Θα επανέλθω στην ε, αναφορά υπαριθμών 30. Εκεί δεν υπάρχει παράβαση του κοινωτικού δικαίου. αλλά όλες οι αναφορές μέχρι 32 πλην τις 30 ε, καλύπτονται. Την 29 την κάλυψα, έτσι. Την 28 φυσικά είναι του κυρίου Κίνγκ, την 31 επίσης και την 32. Τις κάλυψα μαζί, γιατί τα θέματα είναι παρόμοια. Και τώρα θα ήθελα να απαντήσω ε, στο ερώτημα της κυρίας Γουάλης. Με βάση τα όσα ξέρουμε, όντω το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μόνη χώρα που έχει ένα σύστημα α, όπως αυτό που περιγράψετε. Στέλνει το διαβατήριο με το ταχυδρομείο. Σε ορισμένα κράτη-μέλη μπορεί να ε, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα να στείλει το διαβατήριο ε, με το ταχυδρομείο, αλλά μπορεί να πας και ο ίδιος ε, στην κοινότητα. Ε, στο Δημαρχείο, στο Κοινοτικό Γραφείο κτλ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο έτσι γίνεται. Αλλά με βάση το κοινοτικό δίκαιο δεν υπάρχει λεπτομερής διαδικασία για το πώς θα στηθούν οι διαδικασίες, θα το πώς κινηθούν οι διαδικασίες για να διεκπαιρεθούν οι αιτήσει. Και ο κανόνας για τη διαμονή για πέντε χρόνια, ήδη στην έκθεση του Δεκεμβρίου του 2008, ε, για την οδηγία, η Κομισιόν είχε πει ότι αυτό ακριβώ είναι σοβαρή παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Πιστεύουμε ότι είναι αντίθετο με το κοινοτικό δίκαιο λοιπόν αυτό το σημείο και θα αποτελέσει και τμήμα του διαβήματο προ τι Βρετανικέ Αρχέ. Διάβημα που θα οδηγήσει τελικά στη διαδικασία επί παραβάση. Αλλά πάντω ε, έχουμε έρθει σε επαφή με τι Βρετανικέ Αρχέ, έχουμε τη δική του ερμηνεία και την έχουμε γραπτό. Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να αλλάξουν ε, ερμηνεία οι Βρετανικέ Αρχέ. Να πάω τώρα στο σημείο 30 για να κλείσουμε το θέμα με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Ας πάμε και στην τελευταία παρέμβαση που αφορά την αναφορά υπαριθμών 30. Ένα σύντομο ερώτημα για τα πέντε χρόνια. Υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν τον κανόνα του, των πέντε ετών και ποια ερμηνεία δίνουν για αυτόν τον κανόνα, Πώ εφαρμόζουν αυτά τα πέντε χρόνια. Ε, τα πέντε χρόνια όλα μαζί ή πέντε χρόνια από τη στιγμή της εισόδου, όπως κάνουν οι Βρετανοί. Το Βέλγιο ισχύει, στο Βέλγιο ισχύει ο ίδιος κανόνας. Η οδηγία είναι πολύ απλή. Λέει ότι τη πέντε οπω ε, διαμονής χωρίς διακοπή έχεις το βελγιο ισχυει στο βελγιο ισχυει ο ιδιο κανονα μόνιμης άδεια διακοπη εχει το δικαιωμα μονιμης αδεια διαμονή. Το Βέλγιο και οι Βρετανικές αρχές λένε εντάξει, θα πρέπει αυτές, αυτά τα πέντε χρόνια να εντάσσονται στα πλαίσια της οδηγίας. Και εσύ ως Ρουμάνος, ας πούμε, που παρέμεινε στον Ηνωμένο Βασίλειο νόμιμα από το 2003, ας πούμε, λέω, ας πούμε, δεν έμενες μεταξύ του 2003 και 2007 ως πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η, η περίοδός σου ξεκινάει από την 1η Ιανουαρίου 2007 και την 1η Ιανουαρίου 2012 θα έχει συμπληρώσει την πενταετία και θα έχει το δικαίωμα μόνιμης άδειας διαμονής. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν έχετε δικαίωμα εσείς σε Βρετανία να εξαιρείτε ε, το διάστημα της νόμιμης παραμονής πριν ενταχθεί η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό τον όρο ότι το άτομο που διέμενε ε, πληρούσε τις προϋποθέσεις. Εντάξει. Το, κάνει, λοιπόν, το Ηνωμένο Βασίλειο το κάνει και το Βέλγιο. Λοιπόν, ε, ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε τελικές ε, ε, διευκρινήσεις από τις Βρετανικές Αρχές και το ξαναβλέπουμε το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Προχωρούμε, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, με δύο ε, αναφορές, τη 40 και 41, συγγνώμη, 41 και 42 που αφορούν στην Παλαιστίνη, επειδή οι αναφέροντες είναι παρόντες. Ο κύριος David Pegg. <coughs> Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή ε, που μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε την αναφορά μας η οποία ε, θέλει να επαναφέρει τη χρηματοδότηση σε Ισραηλινούς λόγω της κατεδάφισης σπιτιών. Συγκεκριμένα το Ισραήλ, το Ισραήλ έχει κατεδαφίσει πάνω από χίλια σπίτια των Παλαιστινίων η ICAD έχει κατασκευάσει 165 σπίτια και ίσως να θεωρείτε ότι αυτό είναι σταγόνα το ωκεανό από καθαρά ανθρωπιστικούς, ε, ανθρωπιστική σκοπιά πράγματι δεν είναι τίποτα, όμως ε, παράλληλα Πρόκειται και για 165 ε, πράξεις ε, κοινή αντίδρασης Ισραηλινών και Παλαιστινίων που συνεργάζονται και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς ε, κατασκευάζουμε τα σπίτια αυτά ως μια κίνηση καθαρά συμβολική έτσι ώστε να ενθαρρύνουμε την συμμετοχή των Ισραηλινών, των Παλαιστινίων και της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών στο να υπάρξουν νέες συνθήκες για την ειρήνη. Βεβαίω, η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι να στηρίζει τη λύση των δύο κρατών. Όμως ε, οι Ισραηλινοί επιτόπου το παραβιάζουν αυτό, κυρίω ε, κατεδαφίζοντας τα σπίτια των Παλαιστινίων και κατάσχοντας τη γη τους. 60 χρόνια έχουν δείξει ότι δεν μπορεί κανείς να συνεργαστεί με τους Ισραηλινούς. Τώρα η κοινωνία των πολιτών περιμένει από τους Ισραηλινούς να κάνουν κάτι παραπάνω. Ε, πρέπει να αναζητηθεί μια δίκαιη λύση. Και εγώ θέλω να πω ότι το να προσφέρει κανείς τη χρηματοδότηση στην ICAT αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο πρόεδρος Ομπάμα επέλεξε το να σταματήσουν ε, ε, οι παίκτες των επικισμών των Ισραηλινών ότι αυτό είναι μια δίκαιη η λύση. Όμως το Ισραήλ συνεχίζει ε, την κατεδάφιση σπιτιών Παλαιστινίων για να έχει περισσότερο χώρο για τα σπίτια των Ισραηλινών. Και οι δύο αυτές ενέργειες καταδικάστηκαν από τον πρόεδρο Ομπάμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τον στηρίξει τόσο με λόγια όσο και με πράξεις. Και μία σωστή πράξη θα ήταν να προσφερθεί ε, σημαντική οικονομική ενίσχυση στην ICAD. Τα προγράμματα της από το 2002 μέχρι το 2007 χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Φεβρουάριο του 2007, η ΆΕΚΑΤ κατέθεσε προτάσεις έτσι ώστε να αυξηθεί το πρόγραμμα ε, της ανέγερσης σπιτιών, όμως αυτή η αίτησή της απορρίφθηκε. Η Επιτροπή ε, Αξιολόγησης ε, βέβαια είχε δώσει πολύ ψηλή θέση σε αυτή την έκθεση, την είχε κρίνει ιδιαίτερα ικανοποιητική με πολύ υψηλή βαθμολογία. Ο λόγος ε, που δεν εγκρίθηκε τελικά είναι ότι υπάρχουν ε, Παλαιστίνοι που ε, έδωσαν πολύ κακή βαθμολογία στην πρόταση αυτή. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Αν όλα τα κριτήρια πληρούνται, το να αν φαίνεται η πρόταση αυτή ότι συμβαδίζει με την κοινοτική νομοθεσία αν πράγματι προάγει τη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων, ίσω θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι Παλαιστίνοι πολλέ φορές δεν επιθυμούν να έρθουν σε επίσημη συνεργασία με Ισραηλινές οργανώσει, γιατί με τον τρόπο αυτό φοβούνται ότι θα διονυστεί το καθεστώ που επικρατεί. Η εργασία τη ΆΙΚΑ, τα επίσημα και ανεπίσημα, ε, περιλαμβάνει και τη συνεργασία με Παλαιστινίου, και επίσης ε, ε, προσπαθεί να γίνει κατανοητό ότι ε, δεν πρέπει να υπάρχει ε, συνεργασία με τους ε, κατακτητές και γι' αυτόν τον λόγο μέχρι τώρα δεν υπήρχε επίσημη συμμετοχή των Παλαιστινίων. Εμείς όμως θεωρούμε ότι αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος γιατί απορρίφθηκε η πρόταση του Στάινμπερκ η οργάνωση αναζητά ευθύνες για αυτή την αρνητική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει αυτός ο ισχυρισμός εν αυτή η φήμη θέλουμε να ξέρουμε αν πράγματι ισχύει. Η ICAT συνεχίζει το πρόγραμμά της ε, και οι προσπάθειές της στηρίζονται από τους ε, Ισπανούς. Όμως η ICAT αναγκάστηκε να πωλήσει υπαλλήλους, έχει φτάσει μόνο στους τρεις, έκλεισε ένα αποτελεσματικό κέντρο στην Ιερουσαλήμ και έχει περιορίσει κατά πολύ και τις δημοσιεύσεις της. Εμείς γνωρίζουμε ότι η Κομισιόν έχει αξιολογήσει υψηλά τις δραστηριότητες της ICAT και η συμβολή αυτή στις ε, ΜΚΟ για να ευαισθητοποιηθεί η, κοινωνική, η κοινή γνώμη για το Ισραήλ και για τις ε, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινοί. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναθεωρήσει αυτή τη την απόφαση να μην χρηματοδοτήσει την ICAT. Αναγνωρίζουμε ότι ίσως να μην καταστεί δυνατόν να επανεπισκεφθεί η Επιτροπή Επιτόπου της περιοχής αυτές και ίσως στην περίπτωση αυτή να αναζητηθούν άλλες λύσεις για να χρηματοδοτηθεί η ICAT. Ε, από τη μεριά της Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, ε, δεν υπάρχει ε, κάτι με τον οποίο να διαφωνούμε πολιτικά τουλάχιστον με τον αναφέροντα. Στις 15 ε, Ιουνίου οι ε, Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκναν μία δήλωση για την ειρήνη στην ε, Μέση Ανατολή και εκεί αναφέρονται πολλές επιφυλάξεις και ανησυχίες για την κατεδάφιση κατοικιών κυρίως στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Επιφυλάξεις υπάρχουν όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της χρηματοδότησης, κάτι που κοινοποιήσαμε στο παρελθόν στην ICAT. Κοιτάξτε, εμείς δεν χρηματοδοτούμε οργανώσεις, αλλά μέσα από τη συνεργασία για το χρηματοδοτούμε συγκεκριμένα προγράμματα, projects. Έτσι λοιπόν η μη χρηματοδότηση της ICAT δεν σημαίνει μη χρηματοδότηση προγράμματος. Αυτό μπορεί να σας ηχεί γραφειοκρατικό αλλά πρόκειται για μια σημαντική διαφοροποίηση. Εμείς λοιπόν αναφέραμε τους ε, λόγους ε, στους Ισραηλινούς ε, και είπαμε ότι είμαστε ενάντια στην κατεδάφιση των ε, σπιτιών. Βεβαίως και εκτιμούμε τις δραστηριότητές τους και την προσφορά τους στο να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη του Ισραήλ στα προβλήματα που δημιουργούνται. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτό θα μπορέσουμε να το πράξουμε και πάλι στο μέλλον. Τώρα όσον αφορά την οργάνωση την οποία εκπροσωπεί ο κύριος Στάινμπεργκ. Κοιτάξτε, ε, έχουν συμπεριλάβει πολλές, έχουν επιτεθεί σε πάρα πολλές ΜΚΟ και στην ΕΙΚΑΤ για ε, δραστηριότητες που κατά άποψή τους είναι ενάντια στα Ισραηλινά ε, συμφέροντα και στην ΙΚΑΤ. Εμείς λοιπόν χρηματοδοτήσαμε τρία προγράμματα από το 2000 μέχρι το 2005 ύψους 1,1 εκατομμυρίων ευρώ. Νομίζω λοιπόν, γνωρίζουμε με σαφήνεια ότι αυτό το αίτημα του να υπάρχει έλεγχος ε, στις ΜΚΟ ε, αυτό ε, είναι σωστό, αλλά δεν ισχύουν οι υπόλοιποι ισχυρισμοί. Στείλαμε λοιπόν στοιχεία στην ΑΙΚΑΤΕ και στις υπόλοιπες ΜΚΟ και θεωρούμε ότι αν θέλετε μπορούν να σας αποσταλούν τα απαραίτητα στοιχεία. Έχουμε λοιπόν καταστήσει σαφές και στην ΑΙΚΑΤΕ και στην ελεγκτική αρχή ότι δεν ασκήθηκε εξωτερική πίεση στον έλεγχο που διεξήχθη. Η πρόταση θεωρούμε ότι είναι σωστή, αλλά έχουμε ένα αρκετά μικρό ε, κονδύλι για πάρα πολλά προγράμματα τα οποία υποβάλλονται. Και ε, στην περίπτωση αυτά απλά είμαστε αναγκασμένοι να προβούμε σε περικοπή. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Έτσι λοιπόν το γραφείο μας της τεχνικής αρρωγής ε, στην Ιερουσαλήμ ζήτησε να αρθεί αυτός ο ισχυρισμός από την ιστοσελίδα. Το ελέγξαμε βέβαια και δεν έχει συμβεί ακόμα κάτι τέτοιο. Τώρα, όσον αφορά τις, ε, τα αδύναμα στοιχεία της πρότασης της ICAT, νομίζω ότι αυτά προβλήθηκαν σε κάποια άλλη συζήτηση. Τους ζητήσαμε να υποβάλουν καλύτερα τεκμηριωμένες προτάσεις για το μέλλον. Στις τελευταίες συζητήσεις που είχαμε με μία αντιπροσωπεία στο Τελαβίβ καταλήξαμε στο ότι πράγματι υπήρξε μία νέα πρόταση η οποία νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι πράγματι αποτελεί ε, μία δυνατότητα χρηματοδότησης. Σας υπογραμμίζω, εδώ μιλάμε για ε, προτάσεις επιλέξιμες ε, προς χρηματοδότηση. Αυτή λοιπόν την απόφασή μας θα τη λάβουμε μόνο βάσει των προτάσεων που έχουν κατατεθεί. Κύριε Άλτμαν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα τις ερωταποκρίσεις. Ελπίζω να βρείτε λύση, ούτως ώστε το μήνυμα που θα περάσει θα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται πίσω από αυτή την καταπληκτική οργάνωση, τη στηρίζει. Ε, είναι μια θαυμάσια οργάνωση και η επίπτωση του έργου τους σε πολλές χώρες είναι ακριβώς αυτή που περιγράφτηκε. Ε, συνεισφέρουν στο να υπάρξει μια ε, δικοινοτική λύση στην Παλαιστίνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ συχνά λέει το Ισραήλ καταστρέφει, εμείς πληρώνουμε. Πληρώνουμε, πληρώνουμε, πληρώνουμε. Αλλά εδώ πέρα σε εφημερίδες δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τελικά εμείς είμαστε πληρωτές και όχι συμπέκτες. Ε, αλήθεια είναι αυτό. Πληρώνουμε και δεν συμμετέχουμε. Το λένε για αυτό. Ε, το λένε για μα αυτό και είναι αλήθεια. Αυτή η οργάνωση όμω μα καθιστά συμπαίκτε, συμμέτοχου. Είναι πολύ σημαντικό να περάσει αυτό το μήνυμα γιατί είναι πραγματικά μια επικοδομητική οργάνωση. Και ελπίζουμε η όλη υπόθεση να βασίζεται σε μια παρεξήγηση. Ε, εξεπλάγει όταν κατάλαβα ότι το Ισραήλ κατάφερε να σταματήσει η υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ένωση προ αυτή την οργάνωση. Ελπίζω να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία. Η κυρία Γουόλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον συντάκτη της αναφοράς, τον κύριο Πέγκ που μας παρουσίασε την αναφορά. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της ε, Επιτροπής για την πολύ λογική και προσεκτική απάντηση στο δύσκολο αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα χρηματοδότησης όπου πρέπει να δείξουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αποφασίζουμε με κάθε διαφάνεια. Και ότι κάναμε το καταδύναμη. Μία ερώτηση θέλω να σας υποβάλω. Ε, κάποια άλλα προγράμματα προφανώς ε, προτιμήθηκαν. Μήπω θα ήταν δυνατό να μας δώσετε κάποιε ενδείξεις για το ποια ήταν αυτά τα προγράμματα που προτιμήθηκαν. Γιατί νομίζω ότι έτσι θα διασκεδαστούν και οι ανησυχίες που υπάρχουν για το πώς ε, χρηματοδοτούνται τα διάφορα προγράμματα, για το πώς, είναι, πώς έχει η όλη διαδικασία. Όταν ε, για πρώτη φορά διάβασα την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανησύγησα λιγάκι γιατί είδα ότι υπάρχει, η, υπάρχει αλληλογραφία με το NGO Monitor, με αυτή την οργάνωση την Ισραηλινή που παρακολουθεί τις με κυβερνητικές οργανώσεις. Καλό θα ήταν αυτή την αλληλογραφία να τη δει η Επιτροπή Αναφορών για να μας καθησυχάσει. Ε, από τις προφορίες που έχω, συμφωνώ ε, με αυτό που είπατε εσείς, ότι υπάρχουν αυτές οι αναφορές στην ιστοσελίδα Και αυτό δεν βοηθάει την κατάσταση. Σας παρακαλώ, πρόεδρε, μήπως ε, με κάποιο τρόπο μπορούμε να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά για να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Ευχαριστώ. Κύριος Βίγλαν. Κοιτάξτε, ε, πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στο πολιτικό στοιχείο όλης αυτής της υπόθεσης. Ε, εγώ όμω ε, όμως πρέπει να σας πω ότι δεν πρόκειται για αναφορά. Καμία σχέση όλα αυτά που λέγησαν με αναφορά. Εχθές ε, ακούσαμε μια πολύ ωραία παρουσίαση, είτε πρόκειται εδώ για μια λάθος απόφαση, ε, πρόκειται δηλαδή για κακοδιαχείριση και αυτό το θέμα πρέπει να παραπεμφθεί στον διαμεσολαβητή. Εγώ ε, γνωρίζω πάρα πολλές διαδικασίες παρεμφερείς. Αν αρχίσουμε λοιπόν τώρα εδώ να θεωρούμε ως αναφορές τις χρηματοδοτήσεις και τις αναθέσεις σε διαγωνισμούς, τότε φοβάμαι ότι πλέον θα ασχολούμεθα με αναφορές, καμία σχέση όλα αυτά με τη δουλειά μας. Ε, εγώ ε, θεωρώ ότι όταν υπάρχουν λάθος αξιολογήσεις σε χρηματοτήσεις και αναθέσεις διαγωνισμών τότε πρέπει κανείς να καταφύγει σε άλλες αρχές. Υπάρχουν άλλες αρμόδιες αρχές γιατί αν αρχίσουμε εμείς ε, ε, να ασχολούμαστε τέτοιου θέματα τότε ξέρετε που θα καταλήξουμε. Θα καταλήξουμε στον είμαστε εδώ διαγωνισμός ομορφιάς. Να λέμε α αυτό το πρόγραμμα είναι ωραιότερο από το άλλο γιατί το άλλο δεν χρηματοδοτήθηκε. Κοιτάξτε θα κάνουμε ακριβώς αυτό το οποίο οποίο θέλουμε να αποφύγουμε με τη διαδικασία ανάθεσης διαγωνισμών. Ε, αυτό είναι λοιπόν το ένα που θέλω να αναφέρω. Και το άλλο είναι το εξής. Το Κοινοβούλιο αναφέρθηκε με σαφήνεια στα πολιτικής φύσεως θέματα. Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε μια πολιτική επιτροπή η οποία να ενισχύει ε, τα μηνύματα του Κοινοβουλίου που προκύπτουν από άλλες επιτροπές. Θα έπρεπε λοιπόν να ε, ασχοληθούμε περισσότερο με τις ε, ενστάσεις ε, των πολιτών και των οργανώσεων. Τώρα το θέμα το κατά πόσον μπορεί να γίνει παραδεκτή αυτή η αναφορά αυτό αν θέλετε οριακά το συζητάμε αλλά επουδενή δεν είναι αιτιολογημένη και σωστά τεκμηριωμένη το γεγονός ότι ενδεχομένως να λήφθη λάθος απόφαση ας πάνε οι ενδιαφερόμενοι στο διαμεσολαβητή όχι σε εμάς. Και όσον αφορά τώρα του να κρίνονται κατά πόσον οι αναφορές είναι παραδεκτές ή όχι, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να εμπλεκόμεθα σε πολιτική φύσης θέματα, γιατί ξέρετε αλλιώς αν το πράξουμε αυτό ε, πραγματικά θα κάνουμε λάθος δουλειά. Εγώ θεωρώ ότι η αναφορά αυτή δεν πρέπει να κριθεί παραδεκτή. Κύριος άλλη μια φορά. Κυρία, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ. Ε, ναι, είναι αλήθεια, δεν είμαι μέλος της Επιτροπής, αλλά ε, συμμετείχα στην, Παλαιστινιακή, στην Παλαιστινιακή Αντιπροσωπεία στο παρελθόν. Γι' αυτό ε, συμφωνώ με την αναφορά. Και άλλωστε, αυτό φάνηκε και από όλους τους, ε, όλους όσους τοποθετήθηκαν. Ε, κοιτάξτε, πραγματικά, λαμβάνοντα υπόψη αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή το να μην δοθεί ενίσχυση, ε, θα αποτελούσε ένα πολύ άσχημο μήνυμα. Ε, Λαμβάνοντα υπόψη την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, σήμερα περισσότερο από ποτέ ε, είναι η κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο. Το να διακόψουμε τώρα τη χρηματοδότηση. Καταλαβαίνετε ότι ενώ έχουμε τέτοια παραβίαση νομοθεσία ε, και να έχουμε όλους αυτούς τους επικισμούς. Ε, όπως είπε και ένας ε, συνάδελφος, πραγματικά πρόκειται για κάτι ε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σοβαρό. Και αυτό συνδέοντας, και το, συνδέοντα, το συνδέουμε με το γεγονός ότι υπάρχει πίεση επιτόπου από διάφορες οργανώσεις και ότι εδώ δεν πρόκειται ότι εδώ πρόκειται στην ουσία για πρωτοβουλίες ανθρώπων ε, που ε, πραγματικά έχουν δει τους καρπούς της ενίσχυσης στο παρελθόν. Δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ε, και όπως είπε και η κυρία Γόλης, θα ήταν καλό, ίσως όχι ευθύ αμέσω, αλλά θα ήταν καλό να δούμε και ποιες είναι οι άλλες οργανώσεις που πήραν αυτή την ενίσχυση και με βάση ποια κριτήρια. Ε, να δούμε λοιπόν ε, τα πράγματα προς την κατεύθυνση αυτή και τότε να σχηματίσουμε μια πιο ε, ξεκάθαρη και συγκεκριμένη εικόνα της κατάστασης. Γιατί πραγματικά ε, χρειαζόμαστε αυτές τις πραγματικές πληροφορίες. Αυτό είναι σωστό για να μπορέσουμε να το Κυρία Πρόεδρε για να αποφύγουμε τον κίνδυνο ε, εδώ να μπλέξουμε πολλές πτυχές που δεν έχουν ε, ε, σχέση με την καθημερινή μας εργασία. Πραγματικά ζητώ να προσπαθήσουμε να μην αναφερόμαστε σε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία έχουν μια φόρτιση συναισθηματική. Είναι ευαίσθητα, ναι, το δέχομαι, αλλά να ακολουθήσουμε τους κανόνες μας, σύμφωνα με τον κανονισμό μας και σύμφωνα με τις δικές μας αρμοδιότητες πρέπει να αναφερθούμε μόνο σε παραβιάσεις των ευρωπαϊκών των δικαιωμάτων ε, των Ευρωπαίων πολιτών. Να μην ανακατεύουμε τόσα πολλά ζητήματα που βεβαίως συμφωνώ είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, πάρα πολύ σημαντικά. Από ηθική άποψη ε, είναι εξίσου σχετικά με άλλα, αλλά να μην δημιουργούμε την ε, εντύπωση ότι εμείς εδώ ε, τι είμαστε, υπερδικαστές, ε, ιερωμένοι. Μα πρέπει εδώ να καταλάβουμε ποιοι είναι οι δικοί μας κανόνες και οι δικές μας αρμοδιότητες. Εδώ εξετάζουμε τα προβλήματα μόνο τα οποία ε, εμπίπτουν στη δική μας αρμοδιότητα. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση όμως στον κύριο Βοστινάρου Η, η αναφορά κατατίθεται από έναν πολίτη Βρετανό πολίτη της Ευρώπης δηλαδή, εξ ονόματος ενός παραρτήματος στο Ιόρκ μιας, της εκστρατείας ελληνικής στην Παλαιστίνη, αυτής της οργάνωσης. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν έχουμε το δικαίωμα να μην τη λάβουμε υπόψη ως αναφορά. Είναι μία αναφορά. Επομένως, θα πρέπει να τη συζητήσουμε ή να μην τη συζητήσουμε. Δεν συζητάω για το πολιτικό ζήτημα που έθεσε ο κύριος Βίλαντ αλλά δεν είναι μια ερώτηση ενός Ευρωπαίου πολίτη για μια ένωση που έχει παράρτημα στην Ευρώπη. Να προσπαθήσω να απαντήσω. Δεν είμαι ε, δικηγόρος. Αλλά αν υπάρχει παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου θα πρέπει να ε, δοθεί απάντηση, μόνο εφόσον υπάρχει παραβίαση ευρωπαϊκού δικαίου. Και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτούμε αν υπάρχει παραβίαση. Αν ναι, τότε ναι. Ε, εμπίπτει στις δικές μας δραστηριότητες, στις καθημερινές δραστηριότητες. Αλλά να μην κάνουμε τώρα αφαίρετες ερμηνείες. Γιατί τότε θα πέσουμε σε μια τέρμονη ιστορία και νομίζω ότι θα δώσουμε ένα πλήγμα στην έγκλη μας. Ας ασχοληθούμε και ας περιοριστούμε στα προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών και στην παράβαση του ευρωπαϊκού δικαίου και των δικαιωμάτων που απορρέουν από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Κυρία Γουόλης. Ίσως να ε, το βλέπω τα πράγματα υπεραπλουστευμένα, αλλά αναφέρον είναι Ευρωπαίος φορολογούμενος και έχει δικαίωμα να γνωρίζει ε, πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή είχε την ευγένεια να ε, προσφερθεί να μας ε, δείξει τα στοιχεία αυτά, δεχόμαστε ε, την προσφορά. Το μόνο που θα ήθελα να ζητήσω είναι να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιες άλλες οργανώσεις πήραν χρηματοδότηση σε αυτό το γύρο. Γιατί αυτή η πληροφορία θα ήταν χρήσιμη και συγκεκριμένη οργάνωση για την υποβολή νέα αίτηση. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα, αυτό και μόνο ζήτησα. Κυρία Όκα, να προσθέσω το εξή σύμφωνα με τη συνθήκη στο 194 άρθρο είναι παραδεκτή. Μπορώ να σας ε, παραθέσω επίσης οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιοδήποτε φυσικό νομικό πρόσωπο που διαμένει ή έχει την έδρα σε ένα κράτος μέλος έχει το δικαίωμα ε, ε, από μόνο του ή σε αποκοινού με άλλα πρόσωπα να υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα θέμα το οποίο εμπίπτει στη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και που ε, τον αφορά ή την αφορά άμεσα. Και μετά, αν δείτε το, πάτε στον κανονισμό. Και εκεί θα δείτε ότι είναι παραδεκτή. Είναι λεπτή η υπόθεση αυτή, αλλά Πρέπει να το καταλάβουμε. Πρέπει λοιπόν να τη δούμε, ακόμα και αν ε, ε, διατρέχουμε τον κίνδυνο που αναφέρθηκε. Ε, πάντως είναι μέρος της εργασίας μας και νομίζω ότι φυσικά θα πρέπει να δεχτούμε ότι έχουμε την εργασία αυτή. Μπορεί να έχουμε προβλήματα με το Ισραήλ, το ξέρω γιατί εγώ εσωληθεί με το θέμα, το δοκίμασα. Αλλά πάντως έτσι έχουν τα πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Μα είναι μέρος ε, της συνθήκης και μέρος ε, του κανονισμού. Συγγνώμη, δεν ασκώ, δεν είμαι σε κανένα λόμπι, σε καμία ομάδα πίεση, δεν ασκώ πίεση ε, για κανένα. Για να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους. Αυτές οι αμφιβολίες και αυτές οι παρεμβάσεις. Κύριε Βίλαντ. Δεν πρόκειται για το δικαίωμα μιας οργάνωσης ή ενός πολίτη να καταθέσει μία αναφορά. Όμως το θέμα για το οποίο συζητάμε εδώ δεν είναι η πολιτική, το πολιτικό θέμα της οργάνωσης που θέλει να προβάλλει η οργάνωση. Κοιτάξτε, μην αναγκάστε να ανατρέξω στα έγγραφα παλαιότερων συνεδριάσεων, αλλά ε, θα τις άνετα 100 ευρώ για να πω ότι όταν είναι μια οργάνωση η οποία ε, προβάλλει κάτι το οποίο δεν εγκρίνουν οι περισσότεροι και αναφέρει ότι τα πράγματα εκρίθησαν λανθασμένα και οποτεδήποτε αυτό συνέβη στο παρελθόν, μία τέτοια αναφορά πάντα ε, απλώς τελείωνε γραπτά με μια γραπτή απάντηση από τη στιγμή που η Κομισιόν έδινε την πληροφορία ότι ακολουθήθηκε ο νόμος. Εδώ αυτό που παίζει ρόλο είναι κατά πόσον σκόπιμα ή θελημένα ή όχι υπήρχε λάθος αξιολόγηση ε, κατά τη ε, διαδικασία του διαγωνισμού. Αυτή είναι η ένσταση που αναφέρει η συνθήκη και ε, Εάν λοιπόν τώρα έρθει κάποιος και πει ότι ξέρετε εγώ έχω μία αναφορά και το βρίσκω πάρα πολύ λάθος αυτό που αποφάσισε ας πούμε την τελευταία εβδομάδα η Επιτροπή Ελίας θεωρείτε ότι είναι σωστό η Επιτροπή Αναφορών να ασχοληθεί με μία ενδεχομένως λάθος απόφαση της Επιτροπής Ελίας όχι βεβαίως, εμείς δεν είμαστε εδώ επιτροπή για την αξιολόγηση ε, αποφάσεων ε, του Κοινοβουλίου η συγκεκριμένη αυτή υπόθεση δεν είναι δικό μας θέμα. Αυτό που μπορεί να μας αφορά είναι η διαδικασία ανάθεσης. Κοιτάξτε, εγώ πολύ συχνά ασκώ ε, κριτική εις βάρος Κομισιόν, αλλά συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να πω ότι αρκούν οι πληροφορίες που μας έδωσε η Κομισιόν, γιατί, όπως ελέγχθηκε εχθέ, αυτό που ενδιαφέρει είναι η κακοδιαχείριση. Όλα τα υπόλοιπα αφορούν, όπως σας είπα, το διαμεσολαβητή. Εάν λοιπόν ο φορέας πιστεύει ότι στη διαδικασία της ανάθεσης έγινε ένα πολύ σημαντικό λάθος, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να πρέπει να διορθωθεί, τότε ο διαμεσολαβητής μπορεί να επιληφθεί του θέματος. Και εξάλλου, κυρία Γόλης, η διαφάνεια υπάρχει. Μπορεί κανείς ε, να διαβάσει ποιες ε, οργανώσεις επιδοτούνται με ποια ποσά. Αλλά δεν είναι δική μας δουλειά να λέμε ότι «Α, ξέρετε, τώρα ε, χρηματοδοτήθηκαν αυτές οι οργανώσεις, καλύτερα την επόμενη φορά να πάμε στις άλλες». Εγώ επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι αυτή η αναφορά δεν είναι παραδεκτή. Νομίζω ότι τα επιχειρήματα που άκουσα ξεκαθαρίζουν ποια είναι τα όρια των αρμοδιοτήτων μας. Μπορούμε να το δούμε αυτό το θέμα και σε μια άλλη περίσταση. Θα ήθελα να υπενθυμίσω το άρθρο 201 του Κανονισμού για τις Αναφορές, που καθορίζει το δικαίωμα των αναφορών. Για να μην υπάρξει πρόβλημα μετάφρασης, θα το διαβάσω στα αγγλικά. Οποιοδήποτε πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιοδήποτε φυσικό νομικό πρόσωπο που ε, κατοικεί ή έχει το γραφείο του σε ένα κρατό μέλο θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίσει μόνος ή μαζί με άλλους ε, σε οργανώσεις ε, να στείλει μια αναφορά στο Κοινοβούλιο για ένα θέμα που αφορά τον τομέα δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελεία. Μιλάμε για το πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν. Είναι μια ευρεία, λοιπόν, ερμηνεία Επομένως, εντάσσεται σε αυτήν και αυτή η αναφορά. Νομίζω ότι αυτή η αναφορά αφορά αρμοδιότητες ε, της, Επιτροπής Αναφορών, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Συγγνώμη. Επομένως, είναι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο φυσικά. Πρέπει να μην φυστούμε προσπαθειών Θα στείλω λοιπόν αυτή την αναφορά μαζί με ένα σημείωμα ε, στην καθήλυνα αρμόδια επιτροπή που είναι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που ασχολείται με τέτοια θέματα συνήθω. Εντάξει, συμφωνείτε όλοι. Πάμε στο επόμενο σημείο, το οποίο είναι το σημείο 42. Α, τελειώσαμε εγκαίρος. Δεν το είχα καταλάβει. Συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη από το συντάκτη της ε, αναφοράς υπαριθμών 42, γιατί δεν θα καταφέρουμε να συζητήσουμε σήμερα την υπαριθμό 42. Θα πρέπει όλα αυτά τα σημεία να τα παραπέμψουμε στη συνεδρίαση την επόμενη. Επιβεβαιώνω το αίτημα των βουλευτών σε ό,τι αφορά τις αναφορές υπαριθμών, της αναφορές Β, ότι όλες αυτές οι αναφορές θεωρούνται περατωμένες με βάση την συνήθη διαδικασία. Έχουμε δηλαδή στείλει γραπτή απάντηση, έχουν δοθεί απαντήσεις από την Κομισιόν και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τις αναφορές Β, ε, σας προτείνω να κλείσουμε όλες αυτές τις αναφορές. Συμφωνείτε? Ευχαριστώ. Sono 12.30.